Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας. Έχουμε τους προσκεκλημένους μας εδώ και ε, δεν υπάρχει λόγος να τους αφήσουμε να περιμένουν. Παρακαλώ λοιπόν πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη η οποία προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον Γιάνν Φαντερ Χέικ, που αναβάλλεται για το φθινόπωρο και στο συγγνώμη για το λάθος. διερμηνία υπάρχει εκτός της εσθονικής και λιθουανικής γλώσσας. Και θα σας παρακαλέσω να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 3ης και 4ης Μαΐου και της Δευτέρας και 3ης Ιουνίου. Ε, υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις. Όχι, ευχαριστώ. Προχωρούμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Όγκελινγκς. η οποία είναι εδώ ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας, υπεύθυνη για την κοινωνική ενσωμάτωση, και με την κυρία Σαμπίν Λαγουιέλ, που είναι υπουργό Απασχόληση. Όχι. Α, μάλιστα. Α, διατροφικής ασφάλειας. Διατροφικής ασφάλειας και γεωργίας. Δεν ξέρω με ποια σειρά θα λάβετε τον λόγο. Η κυρία Άουγκελίνγκ, φαντάζομαι. Ici, euh, le rapport. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Βέβαια έχουμε να συστήσουμε την έκθεση της κυρίας Γκροστέτ, το, τη δέσμη μέτρων ε, για τα φαρμακευτικά, την ενημέρωση του καταναλωτή που μας απασχόλησε πολύ, την έκθεση της κυρίας Λιωτάχη για τα νέα τρόφιμα, για την οποία δουλέψαμε πολύ σκληρά. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σας ακούμε. Κύριε Όγκελεγξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, κυρίες και κύριοι, η Βελγική Προεδρία αποφάσισε να ε, οργανώσει την πρώτη της άτυπη συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου για τα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα λοιπόν το οποίο μας απασχόλησε. Θα ήθελα να σας δώσω στοιχεία από τις συστήσεις μας καταρχάς είχαμε συζήτηση για τον καρκίνο. Ξέρω ότι σας έχει υποσχολήσει πολύ. Πάνω από 3.200.000 Ευρωπαίοι πέφτουν θύματα της επάρατης νόσου κάθε χρόνο με υψηλά ακόμη δυστυχώς ποσοστά θνησιμότητας. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει λοιπόν, συζητήσαμε στο Συμβούλιο, δεδομένου ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προταθεί, πραγματοποιηθεί, υλοποιηθεί δράσεις ε, για τον καρκίνο, νέα πρόταση δράσης, κοινή δράσης από την Επιτροπή. Από το άτυπο Συμβούλιο λοιπόν αυτό που προκύπτει ως αποτέλεσμα είναι πως τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους συμπράττουν στην κοινή δράση κάποιοι Μάλιστα, ακολούθησαν εκ των υστέρων ε, την άτυπη συνεδρίαση, το άτυπο συμβούλιο, να έχουν όλα τα κράτη ένα σχέδιο δράσης για τον καρκίνο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσω των δυνατόν καλύτερα ποσοστά έγκαιρης διάγνωσης για τα ε, για τις μορφές τουλάχιστον εκείνες καρκίνου όπου η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να ε, σημάνει και μεγάλη ε, διαφορά ως προς την εξέλιξη της νόσου, όπως σε παραδείγμα στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Το ίδιο μας απασχόλησε στο άτυπο αυτό Συμβούλιο Υπουργών Υγείας το θέμα του, ε, της νέας γρήπης H1N1 που μας είχε απασχολήσει εδώ και καιρό όπως γνωρίζετε με το, με το κίνδυνο μιας πανδημίας που είχε προεξαγγελθεί. Παρακολουθήσαμε τους τελευταίους μήνες την εξέλιξη αυτή σε πραγματικό χρόνο και όταν όπως το Βέλγιο είχε ζητήσει Φερρυπίν μεταξύ άλλων κρατών. Γινόταν λόγος για μια κοινή διαχείριση των παραγγελιών και της αποθήκευσης των εμβολίων 21 εκ των 27 κρατών αντιδρούσαν. Είδαμε εντωμεταξύ, όπως είπα σε πραγματικό χρόνο, την εξέλιξη της πανδημίας και στο άτυπο συμβούλιο είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι δεν εκφράζονται πλέον αντιρρήσεις σε, ε, στην δυνατότητα να εργαστούμε από κοινού για την ε, διαπραγμάτευση Φερρυπίν και την ε, διατύπωση ε, Ενό προγράμματο για τα νέα εμβόλια και τα σχετικά βέβαια θα μα τα προτείνει στι αρχέ του φθινοπόρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε ασφαλώ σε λίγο. Αλλά πάντως πρέπει να σημειώσω ότι υπήρχαν λόγω του κατακαιρματισμού της διαχείριση της ε, πανδημίας ε, της γρηπη h H1N1 πολλές, πολλές πολλες δυσκολιε Επίσης το Υγειονομικό Συμβούλιο του οποίου η εντολή ε, εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου και πρέπει να δούμε ε, πώς θα συνεχίσει τις εργασίες του. Μας απασχόλησε στο Αττικό Συμβούλιο. Ε, άλλα σχετικά σημαντικά ζητήματα νομοθεσίες όσον αφορά τη δημόσια υγεία μας απασχόλησαν και ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται να πραγματοποιήσουμε έξι δεσκέψεις ανώτατου επίπεδου, μία στις 20 Οκτωβρίου για τις χρόνιες νόσους, σε αρχές Σεπτεμβρίου για το υγειονομικό προσωπικό, όπου ασφαλώς θα τα γνωρίζετε εσείς σε κάθε κράτος μέλος σχεδόν παρουσιάζονται λήψεις, προβλήματα προς την πρόσβαση, στο επάγγελμα ποιότητας κτλ. Επίσης υψηλού επίπεδου διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί και το, Σεπτέμβριο και για θέματα διατροφής, τέταρτη διάσκεψη 20 3-24 Σεπτεμβρίου για την καινοτομία ε, και την παραγωγή στον χώρο του φαρμάκου, ιδιαίτερα για το θέμα της πρόσβασης του ασθενούς σε φάρμακα, σε, περίπτωση, σε φάρμακα καινοτόμα, σε περίπτωση ορφανών ασθενειών, νόσων. Διάσκεψη θα γίνει και ως προς την άνοια και δει την ε, νόσο του Αλτσχάιμερ ε, νέα δεδομένα, συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κτλ. Και μία διάσκεψη, μία και 2 Οκτωβρίου, για την κατάρτιση τη σχετική με την εφημερία των ζώων. Αυτές είναι οι προτάσεις του Συμβουλίου για το Σεπτέμβριο, ακόμα για το φθινόπωρο, ως προς τις διασκέψεις και τώρα περνώ στα νομοθετικά μέτρα με πρώτα τα φάρμακα, όπου θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαίρετη συνεργασία μας που μας επέτρεψε, πιστεύω, να καταλήξουμε στην οδηγία για την φάρμακο επαγρύπνηση. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι η κοινή μας δουλειά, η συνεργασία μας και μάλιστα πρέπει να πω ότι αποτελεί και ε, καλό ιονό για το μέλλον, για τα φαρμακευτικά μια δεύτερη πρόταση που ασφαλώς γνωρίζετε πολύ καλά είναι η πρόταση οδηγίας που έχουμε στο Συμβούλιο για τα, παρα, ε, για τα πειρατικά ή παραποιημένα φάρμακα. Παρακολούθησα τις σημαντικές εργασίες της Επιτροπής πρέπει να βρούμε λύσεις ε, ως προς τις διαφορές οι οποίες αφορούν, ε, χαρακτηρίζουν τους ορισμούς, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας. τις παράλληλες ε, παραγωγές. Βέβαια, έχετε εσείς ξεκινήσει ένα νέο πεδίο δράσης με, το, με την πώληση μέσω του ίντερνετ ένα πεδίο πολύ σημαντικό πιστεύω, καθώς 60% των φαρμάκων που πολλούνται στο ίντερνετ είναι παραποιημένα, είναι αντίγραφα και ασφαλώς ε, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί αυτή η αυτή η περίπτωση, αυτό το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν ε, να βοηθήσουμε ώστε να καταλήξουμε σε ε, αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό, το φθινόπωρο μαζί με, τους, ε, μαζί με το Συμβούλιο γιατί πολύ συχνά έχουμε προβλήματα ε, ως προς την αντιγραφή των φαρμάκων. Η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε ως προς το κείμενο της Επιτροπής που είχε αρχικά αυτή την ιδιαιτερότητα ότι δηλαδή ε, ε, κατάφερε να το καταπολεμήσουν οι πάντες. Το Συμβούλιο λοιπόν ότι θέλει να συζητήσει την πρόταση αυτή. Στο άτυπο Συμβούλιο επανέφερα το θέμα, το ξανασυζήτησα με τους συναδέλφους και βλέπω ότι υπάρχει διάθεση τουλάχιστον να το συζητήσουν. Και πλέον πρέπει με βάση αυτή την ε, συζήτηση, αυτή τη βούληση αν θέλετε, να δούμε εάν μπορούμε να εξασφαλίσουμε συμφωνία ο Επίτροπος Δαγή που ήταν παρόν κατέγραψε τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσει προκειμένου να προσαρμόσει το κείμενο βέβαια και στις προτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ανακοίνωση νομίζω έχει ήδη προταθεί στο Κοινοβούλιο να μην ε, ανακληθεί η ανακοίνωση αλλά να αναλυφθούν να ληφθούν υπόψη τα, οι παρατηρήσεις του ε, Κοινοβουλίου. Αυτά για τα φαρμακευτικά. Επίσης έχουμε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο κείμενο των ε, υπερσυνοριακών υπηρεσιών. Ένα κείμενο το οποίο έχει να κάνει βέβαια πάνω απ' όλα με τα συμφέροντα των ασθενών. Ξέρετε ότι χρειάστηκε να εναλλαχθούν στην Προεδρία ε, τέσσερις προεδρίες μέχρι να φτάσουμε τον προηγούμενο Ιούνιο σε μια συμφωνία. Το κείμενο που αποτέλεσε αντικείμενο πολιτικής συμφωνίας βέβαια παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτό που θέλατε. Η βούλησή μου και πάλι είναι να εργαστούμε α, στενά, να συνεργαστούμε στενά μαζί με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή και έχοντας ε, παρακολουθήσει βέβαια τις εργασίες του Κοινοβουλίου μπορώ να σας πω ότι δεν είναι δεδομένες οι ε, δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες για την υγεία για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα βεβαίως θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι κάθε κρατος μέλος προσπαθεί να έχει επαρκή ε, χρηματοδότηση του εθνικού συστήματος ε, προσφοράς υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι κάτι, η χρηματοδότηση δηλαδή και η παροχή των υπηρεσιών έχουν και οι δύο ως κύριο γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς. Άρα πρέπει και αυτά να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Άλλα δύο θέματα είναι η ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τα τρόφιμα. Το Κοινοβουλίο σας μόλις υιοθέτησε την έκθεση από τρεις εβδομάδες και ε, σας συγχαίρω εκ μέρους Συμβουλίου. Το Δεκέμβριο ε, ελπίζουμε σε μια πολιτική συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου για να προχωρήσουμε στη δεύτερη ε, ανάγνωση χωρίς... Ε, να υπάρχει συμφωνία σε όλα τα θέματα, επί παραδείγματι το ζήτημα της σήμανσης, ε, αλλά και το ζήτημα της σήμανσης για την προέλευση, το ζήτημα γενικότερα της ενημέρωσης, της αναγραφής για τα αλκοολούχα ποτά, οι εθνικές ε, ε λύσεις και οι διατροφική σήμανση. Μετά το θέμα του novel food, τα νέα τρόφιμα, όπου πρόσφατα σε 7 Ιουλίου λάβατε σαφέστατες ε, αποφάσεις και επιλογές τους προς τα κλωνοποιημένα ζώα, τρόφιμα προερχόμενα από κλωνοποιημένα ζώα, μεγάλη απόκληση μεταξύ των προτάσεων της Επιτροπής και αυτών του Κοινοβουλίου. Επίσης από το Συμβούλιο θα πρέπει ασφαλώς να τοποθετηθούμε και βλέπουμε στον ορίζοντα τη διαδικασία της συνδιαλλαγής για τις προσεχείς εβδομάδες. Βεβαίως και αποκλίνουν οι απόψεις πλην όμως. Έχουμε συνέντευξη πιστεύω και η ΜΕΝ και η ΔΕ ότι χωρίς την επίτευξη συμφωνίας η διάθεση στην εμπόριο των κλωνοποιημένων προϊόντων πραγματοποιείται μέρα με τη μέρα και προχωρεί. Άρα το laissez δεν είναι λύση και θα πρέπει πάντως να εργαστούμε και μάλιστα πολύ γρήγορα για να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό σε μια συμφωνία μεταξύ μας. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, για τα όσα θα μας απασχολήσουν στις επόμενες εβδομάδες. Κυρία Υπουργέ και Πρόεδρε του Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας, τα ανοίγματα σε αυτές τις παρατηρήσεις που καταδεικνύουν ότι το έργο σας θα είναι αξιόλογο και ιδίω όσον αφορά το τελευταίο σημείο για την κλωνοποίηση θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο έχει μια κρυστάλλινη σταθερή θέση και θέλουμε να επανέλθουμε και στην συνδιαλλαγή πρόκειται πολλά να γίνουν και τώρα να δώσουμε την σκητάλη στην κυρία Υπουργό την κυρία Λαριέλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όσον αφορά τα κτηνιατρικά και τα φυτοϊγειονομικά και διατροφική ασφάλεια, εμείς θέλουμε να προωθήσουμε κάποιες πολιτικές συνέπειες, διαχείριση κινδύνου, ό,τι έχει σχέση με την παγκοσμιοποίηση συναλλαγές, ανταλλαγές, κλίμα, αλλαγές του κλίματος, συγκέντρωση κτηνοτροφικής δραστηριότητας και όλα αυτά επιβάλλουν το να υπάρχει μια πολιτική πρόληψης ανάλυσης κινδύνου η οποία θα συνεχιστεί ε, υπό όρους που θα είναι συμφέροντες εις τους κτηνοτρόφους και γεωργούς. Να δούμε επομένως τι γίνεται αυτή η κρίση του 2007 που μας έδειξε ότι οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών έχουν επιπτώσεις εις το κόστος των ειδών διατροφής και κτηνοτροφής. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε έλλειμμα όσον αφορά την φυτική πρωτεΐνη το έχουμε τα εξή. Πρώτα απ' όλα το χάρτη πορεία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια αξιολόγηση όσον αφορά την εγκεφαλοπάθεια των βοηδών για την περίοδο 2010-2015 γιατί δεν θα πρέπει να τεθεί εν κινδύνο δημοσία υγεία. Και όταν έχουμε κάποιο είδους ατυχήματα θα πρέπει να μπορούμε σε περίοδους τέτοιων ξαφνικών κρίσεων να υπάρχει άμεση αντίδραση και μέχρι ότου ε, απομακρυνθεί ο κίνδυνο, θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε τι αξιολόγηση έχει η Κομισιόν, ούτω ώστε να έχουμε συστήματα αξιολόγηση κινδύνου σε κάθε φάση. Επίσης θα πρέπει να απλουστεύσουμε κάποιες διαδικασίες για την διατροφική ασφάλεια και κινδύνους υγείας. Δεύτερον, χρηματοδότηση της στρατηγικής για την υγεία των ζώων και σας παραπέμπω στο Συμβούλιο που θα συζητήσει, θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου, ούτω ώστε ε, και όσον αφορά την, τα φυτογειονομικά, ο ε, Επίτροπος Νταλή πρόκειται να παρουσιάσει ε, σχετική αναφορά έκθεση. Αυτό θα γίνει και επίσης θα σας μιλήσει και εδώ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δύσκολο θέμα, έχει πολλές πλευρές, καλλιέργεια, αδειοδότηση και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι το Συμβούλιο της Γεωργίας ε, βεβαίως και θα εμπλακεί στο θέμα διότι ε, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει επίπτωση στο περιβάλλον θα έχουμε μια τέτοια ένα τέτοιο συσχετισμό ε, με τα προβλήματα της γεωργίας γιατί ακριβώς το θέμα μας εδώ είναι το πώς αυτοί οι οργανισμοί ε, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις καλλιέργειες. Επομένως θα έχουμε την ε, εισήγηση Νταλή και θέλει η Προεδρία μας να επεξεργαστεί περαιτέρω το θέμα. Πρώτα-πρώτα έχουμε τον Οκτώβριο Συμβούλιο αυτήν την διάσκεψη όπου βεβαίως και θα είστε προσκεκλημένοι. Αυτό το συμπόσιο όσον αφορά τον ρόλο της επιστήμης για την διατροφική πολιτική και θέματα θα είναι επιστήμη πρώτον και αλήθεια. Επιστήμη και δημοκρατία. Είναι δυνατόν κανείς να αναθέσει να, στους επιστήμονες να αποφασίζουν. Και τρίτον, η αρχή της πρόληψης, κάτι το οποίο ισχύει κάτι εξοχήν για το τι θα γίνει με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, δεν μακρηγορώ, αλλά ευχαριστώ να απαντήσω στις τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Ναι, για αυτά τα θέματα βεβαίως και με το θέμα της καλλιέργειας όσον αφορά τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Ε, ça ne veut pas dire que c'est la seule considération à prendre en compte, mais bien sûr que ça concerne l'agriculture. Πρόεδρος. Για να δώσουμε τώρα τις κοιτάλεις στους ε, συναδέλφους. Ε, όχι πάνω από πέντε. Δυο δυ, λεπτά. Ο καθένας, κύριε Γκροστέτη, πρώτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ειδικότερα κάτι που είναι υπεύθυνοι για την υγεία. Μας δώσατε κάποιες ενδείξεις όσον αφορά το τι θέλετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας σας. Δεν σε εκπλήσει ότι ως εισηγήτρια όσον αφορά τα δικαιώματα των ασθενών για τη διασυνοριακή περίθαλψη. Δεν σε εκπλήσει λέγω ότι επιμένω ως ιδιαίτερος επί των θεμάτων αυτών λέγοντά σας ότι πραγματικά βασίζομαι επί της Βελγικής Προεδρίας Επιτρέψε μου να χαιρετήσω εξάλλου τις καλές σχέσεις που έχουμε με τις υπηρεσίες σας για να μας δίνουν αυτές οι υπηρεσίες όλες τις καλές πιθανότητες να καταλήξουν πολιτική συμφωνία προεδρίας σας διότι όπως είπατε χρειάστηκαν τέσσερις διεδοχικές προεδρίες για να καταλήξουμε κάπου χάρη στην Ισπανική ε, Προεδρία σε μια συμφωνία γνωρίζοντας ότι είναι πρώτη φορά που έχουμε μια θέση του Συμβουλίου η οποία δεν ε, εφαρμόζεται στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και καθήκον μας είναι να βρούμε μέσα προσεγγίσεως ούτως ώστε να βρούμε πραγματικά μια λύση διότι αυτή η οδηγία αναμένεται από τους ασθενείς ε, περιέχει κάποιες αβεβαιότητες όσον αφορά την επιστοφή των εξόδων, την προσβασιμότητα στην περίθαλψη, τι γίνεται σε διασυνορικό επίπεδο επί της κλινικής παρακολουθήσεως, όλα αυτά που δεν θέλουμε συστηματικά να είναι προβλήματα. Και επενθυμίζω ότι αυτή η οδηγία δεν έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή περίθαλψη αυτή κάθε αυτή, αλλά να την καθιστά δυνατή να είναι ασφαλής, ποιοτική και χρήσιμη. Η Ισπανική Προεδρία, όπως είπα, κατέληξε σε κάποια συμφωνία, μας οδήγησε συμφωνία. Βασίζομαι στην καλύτερη δυνατή συμφωνία με τη Βελική Προεδρία για να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας, διότι είναι σημαντικό να ωφεληθούν οι συμπολίτες μας, οι ασθενείς, να ωφεληθούν από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σεβόμενοι βέβαια τις εθνικές αρμοδιότητες όσον αφορά την οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών ε, περίθαλψης. Θα πρέπει να σεβαστούμε βέβαια την αρχή της επικουρικότητας. Μίλησα εκ των προτέρων αντιδότηση. Έχουν πολλά ερωτηματικά όσον αφορά την επιστροφή των χρημάτων, τον ορισμό των, των υπηρεσιών περίθαλψης. Πολλά ερωτήματα, κυρία Υπουργέ. Τι περιμένω από εσά. Περιμένω να μου πείτε ότι είσαστε εξίσου αποφασιστικοί όπως και εγώ, ώστε να καταλήξετε σε μια πρόταση, σε μια συμφωνία που να ικανοποιεί πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά και επιτέλους να βρούμε τη λύση. Μιλήσατε για τα παραποιημένα φάρμακα. Ανησυχώ, διότι θεωρώ ότι κολλησιεργούμε. Κολλησιεργούμε ενώ πρόκειται περί εγκληματικότητος και Περιμένουμε το κείμενο τόσο καιρό πια και θα ήταν λυπηρόν να χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Και για να μην μακρηγορώ, ας ολοκληρώσω. Αναφερόμενοι στην αναθεώρηση οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της υγείας πάντα, να σε επιστήσω την προσοχή επί των διακυβευομένων αυτής της αναθεωρήσεως. Διακυβευόμενα για τους ασθενείς, για την ασφάλεια της περίθαλψης που θα πρέπει να είναι να έχει προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μεγάλε διαβουλεύσει επ' αυτού. Θα πρέπει να ακούσουμε του ενδιαφερόμενου κύκλου, κυρίω του ιατρού, ούτω ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση στον αφορά την περίθαλψη που παρέχεται στου ασθενεί. Θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, να μου πείτε κάτι όσον αυτό το θέμα, βασικό θέμα κινητικότητα των ασθενών. Εάν είσαστε δεσμευμένοι να φτάσετε εις βάθος όσον αφορά τα θέματα αυτά και να καταλήξετε σε κάποια συμφωνία μαζί μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίλμοτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Όγκελιξ, το πρόγραμμα της Βελικής Προεδρίας, αυτή η προετοιμασία και ο συντονισμός για την σύμβαση, για τον έλεγχο καπνού, για τη σύμβαση αυτή που θα γίνει το Νοέμβριο, έχει προτεραιότητα. Μπορείτε να επεκταθείτε. Κυρίως για το πρωτόκολλο για το παράνομο εμπόριο ξέρουμε αποτελεσματικός τρόπος να μειώσει, μειωθεί η κατανάλωση καπνού είναι να αυξήσει κανείς τις τιμές μέσω αυξήσεως της φορολογήσεως. Θα έχουμε πραγματικά συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση. Θα υποστηρίσετε σύστημα ανείχνευσης προϊόντων καπνού. Απαγορευτεί η πώληση διαδικτύου και ε, εκ της αποστάσεως πώληση που φοροδιαφεύγει είναι και το θέμα της πολύ χαμηλής φορολόγησης των τσιγάρων σε κάποια κράτη-μέλη. Θα το εξετάσετε αυτό επί της Προεδρίας σας. Και τέλος, με θλίψη γνωρίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μιλούμε με μεγάλο κύρος επί των θεμάτων αυτών, διότι ακόμα δεν έχουμε τακτοποιήσει τα των οίκων μας τακτικά παραβιάζουν την απαγόρευση καπνίσματος οι ευρωβουλευτές στους χώρους του Κοινοβουλίου παρά το ότι έχουν φτιαχτεί ειδικέ καμπίνε για να καπνίζουν και ίσω ε, πρέπει να το εξετάσει η πρόεδρος επιτροπή μα. Δεν τίθεται εν κινδύνο μόνο η ζωή του προσωπικού ε, του Κοινοβουλίου, κυρίω των μελών του μπαρ, του προσωπικού του μπαρ, αλλά αμαυρώνεται ε, κάπως η εικόνα Επιτροπής που θέλει να κινηθεί όσον αφορά την απαγόρευση του, του καπνίσματος και τον περιορισμό του καπνίσματο και του εμπορίου καπνού. Ευχαριστώ κυρία Ντελβού, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις να θέσω προς την κυρία Όλκε Λίνξ. Το πρώτο ερώτημα αφορά την γρήπη ή τα 1-1. Αναφερθήκατε σε αυτή την πανδημία και τη δυνατότητα να αντιταχθούμε σε δεχόμενη νέα πανδημία. Συλλογικά και συντονισμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει προτάσεις μέχρι το φθινόπωρο και να υποβάλει πρόσκληση βολή ενδιαφέροντος για τα εμβόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει οι όροι της προτάσεως να διαφωτιστούν όπως και η διαχείριση των αποθεμάτων. Θα ήθελα ξέρω ποια είναι η πρότασή σας επ' αυτών των δύο συγκεκριμένων θεμάτων. Άλλο ερώτημα που αφορά την οδηγία για τη συνοριακή περίθαλψη στην τομέα τη υγείας. Το Συμβούλιο πράγματι κατέληξε σε συμβιβασμό επί της οδηγίας. Ο στόχο, ο επιδιωκόμενος από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν να δοθεί σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στου ασθενεί αλλά αληθεύει και το είπε και υπάρχει και το συνέστημα, του συμβαστικό κείμενο δεν καλύπτει όλες τις νομικές αβεβαιότητες και θα ήθελα να θέσω και εγώ το ερώτημα. Ως υπουργό Υγείας, μέλος του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ, έχετε τη φιλοδοξία να α, καλυφθούν οι νομικές αβεβαιότητες από το κείμενο μέσω τροποποίησεώς του και αν ναι, Μετά, μιλήσατε για τον καρκίνο. Εγώ θέλω να μιλήσω για άλλη μαστίγα. Το AIDS. Ξέρουμε ότι η πρόληψη και πρώιμος εντοπισμός είναι κάτι σημαντικό. Και τίθεται θέματα επικουρικότητας, σαφέ αυτό. Αλλά η Ευρώπη μπορεί να δώσει κάποια όθηση. Ερώτημα. Η Βελική Προεδρία έχει φιλοδοξία να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συντονίσουν καλύτερα αυτές τις προσπάθειες και να εστιάσουν καλύτερα τις προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την έγκαιρη ε, διάγνωση του AIDS, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ενδεχόμενη θεραπεία και να γίνεται καλύτερο χειρισμός τη ασθένειας. Ευχαριστώ. Φρέντερικ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις υπουργούς μας για την αρχική τους παρουσίαση και όλα τα ερωτήματα που ήδη αναφέρθηκαν ακροθυγώς και τα ζητήματα που εθίγησαν συνοπτικώς, αλλά είναι ικανός του παιχνιδιού βλέπετε να ευχαριστήσω την κυρία Βίλμοτ για την παρουσίασή της που επιτρέπει να μην αναφερθώ στο καπνό. Την υποστηρίζω πλήρω σε αυτά που μας έθεσε και τα ερωτήματα που έθεσε. Από εκεί και πέρα να ζητήσω την ενθάρρυνση της κυρίας Όγκελινγκ. Τον, Ιούνιο τον Ιούνιο το πακέτο για την δωρεά οργάνων και σχέδιο δράσεω ετοιμάζεται με έξοχη συνεργασία τριών προεδριών που συνεργάστηκαν εντατικά γι' αυτό. Είναι ένα πακέτο που ψηφίστηκε, αλλά θα πρέπει να προσγειωθεί το ταχύτερο δυνατόν. ομαλή ανομαλή προσγειωσή του και εν ονόματι των δεκάδων χιλιάδων ασθενών που περιμένουν δωρεά οργάνων, καλό θα ήταν να είναι ομαλή αυτή η προσγείωση τελικά αυτού του πακέτου. Ήθελα να το αναφέρω και αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Λαγουέλ. Άκουσα ότι στα σεμινάρια της διασκέψης που θα λάβουν χώρα δύο σεμινάρια και δύο παρουσιάσεις για τελώς ανεξάρτητα θέματα. Ανεξαρτησία της εμπειρογνωμοσύνης, περίθαλψη, μη περίθαλψη, ε, έλλειψη περίθαλψης και αντιμετώπισης της, ε, νέα, του νέου της γρήπης. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και αφορά όλα τα ζητήματα που συζητούμε εμείς. Καμιά φορά τα συζητάμε καλά, καμιά φορά λιγότερο καλά. Αναφερθήκαμε σε κάπως καυτά θέματα του τροπημένους οργανισμούς. Σας πάμε τώρα στην ανατεχνολογία. Και αυτό που αφορά όλα τα ζητήματα, διαχέει όλα τα ζητήματα, πολλέ ευθύνε, πολλέ αρμοδιότητε όσον αφορά την ανατεχνολογία και τι χρήσει τη ανατεχνολογία. Μεγάλο θέμα. Και οικονομικό και επιστημονικό, με εξαιρετικά ποικιλόμορφε εφαρμογέ σε πολλού κανονισμού και Οδηγίε ψηφίσαμε τεχνολογία και στα καλλιντικά, το θυμάται Ντάγμαρ, ζητήσαμε να αναφέρονται αν περιέχονται προϊόντα ανατεχνολογία και τι γίνεται με τη χρήση προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα κλπ. Το θέμα τη ανατεχνολογία είναι πολύ σημαντικό βεβαίω στην οδηγία. Ε, διάβασα προσεκτικά νομίζω το πρόγραμμα της Προεδρίας. Δεν βλέπω, δεν βλέπω το θέμα να αναφέρεται. Δεν λέω ξαφνικά βεβαίως να το ξαναβάλουμε στο χρονοδιάγραμμα, αλλά ξέρω ότι η Προεδρία εργάζεται συντονισμένα και συντονίστηκε με την Ουγγαρία. Να αποφύγουμε την έλλειψη συζητήσεως για την τεχνολογία και για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Λόγω ελλείψεως γνώσεως να μην ε, δίνουμε εικόνα διαβολική σε κάποια προϊόντα. Επιστήμη αλήθεια ποια είναι και η τεχνολογία; Η Βερική Προεδρία μπορεί να συνεργαστεί με την Ουγγρική Προεδρία ούτω ώστε να ξανασυνδέσει αυτό το βαγόνι στο τρένο των εργασιών της. Ενδιαφέρεται πολύ κοινή γνώμη. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος. Ο Νικόλα Σαρκοζή στη Γαλλία δεσμεύτηκε στα πλαίσια του περιβάλλοντος να συζητήσουμε διάφορα θέματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συζητήσουμε όλα αυτά. Περιμένω να ακούσω τι έχετε να πείτε όσον αφορά τα αντικειμενόμενα. Σα περιμένω. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ, Παγνιού. Κυρία Αναπληρώτρια Πρωθυπουργέ, αγαπητοί φίλοι, με χαρά σας ξαναβλέπω εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να θέσω μια σειρά ερωτήσεων και παρατηρήσεων για τη Βελγική Προεδρία και το προσεχές εξάμεινο. Μιλήσατε για την πρόληψη, για τον καρκίνο. Είχαμε μια έκθεση πρωτοβουλία που υιοθετήθηκε. Εγώ ήμουνα εισηγητή εκ ομάδα μου για την έκθεση αυτή. Ο κύριο Πέτερλε είχε την ε, ε, έκθεση την ίδια. Η Βελγική Προεδρία ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ε, προωθήσει μια οδηγία για την πολύ σημαντική αυτή οδηγία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτρέψει εναρμόνιση των πολιτικών πρόληψης και καταπολέμηση του καρκίνου. Για την ε, γρήπη H1N1, τις τελευταίες εβδομάδες στο Κοινοβούλιο με τον κύριο Λεπάζ, Λεπαζή, τον υποφαινόμενο που είχαμε ζητήσει μια επιτροπή έρευνας, διερεύνησης υπόθεσης, ε, αγωνιστήκαμε, το Προεδρείο του Κοινοβουλίου δεν δέχτηκε την Ερευνητική Επιτροπή και, και τη βέβαια ε, ε, υποκλίνομαι σε αυτή την απόφαση του Προεδρείου που ήταν και πλειοψηφική, θεωρώ ότι ήταν εσφαλμένη, διότι εν ώψη προληπτικής δράσεως σε περίπτωση άλλων ε, πανδημιών που θα, μας, ε, θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και μιλήσατε εσείς για πανδημία, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν πανδημία, ήταν επιδημία. Πολύ λιγότερο έντονη, πολύ μικρότερη ένταση από ότι η εποχιακή, εποχιακή επιδημία της γρήπης που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει στους επόμενους μήνες η Βελγική Προεδρία να εξασφαλίσει την λήψη των διατάξεων εκείνων που θα επιτρέπουν να αναπτυχθούν οι προληπτικές εκείνες αρχές, οι αρχές της πρόληψης και οι, τα μέτρα, τα προληπτικά που θα πρέπει να έχουμε στη θέσή μας για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν. Το Alzheimer's επίσης που αναφέρατε είναι μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες της εποχής και ως προς την ε, ε, διάσταση του ε, προσδόκιμου ζωής, αλλά και συγκεκριμένα μέσα στα κράτη-μέλη βλέπουμε μεγάλη έκταση της νόσου του Αλτσχάιμερ και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να την καταπολεμήσουμε. προσλαμβάνω και μεγαλύτερες διαστάσεις. Τέταρτον, και στο συγγνώμη από την κόρη που μακρηγορώ, αλλά θα συντομεύω, οι υπερσυνοριακές υπηρεσίες. Με τον Λεκλέρ, τον Ντεμότ και την Μαχτίνο Ομπρί είμαστε ε, συμπρόεδροι της μεγάλης αυτής περιφέρειας Λίλ, Κουρτρέ, Τουρνέ και βλέπουμε ακριβώς το φαινόμενο αυτό της διασυνοριακής ε, ε, προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στις οδοντιατρικές υπηρεσίες βλέπουμε μεγάλη άνθηση του φαινομένου αυτού και άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στη ρυθμισή του. Επίσης, ε, ναι, αναζητούμε συμβιβαστικές λύσεις στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, της σχετικής με τη διαφήμιση του φαρμάκου και την ενημέρωση του ασθενούς στην Ευρώπη. Καλό όμως ήταν επίσης το Συμβούλιο, η Βελγική Προεδρία, να μας δώσει τη δική της αίσθηση για το θέμα αυτό η Πρόεδρος. Κυρίες Υπουργοί, έχετε αρκετές ερωτήσεις ε, λάβει. Εγώ θα συμφωνήσω με την Φρεντερίκ Ρίς και τον Ζιλ Παρνιό στις παρατηρήσεις τους ως προς το εμβόλιο της γρήπης H1N1 αφενός και το ζήτημα της ε, εξειδίκευσης. Ένα πρόβλημα το οποίο επανέρχεται όπως και αυτό της εμπιστοσύνης που ε, αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τους ε, ειδικού που έρχονται να μας δώσουν κάποιες γνώσεις πραγματογνωμοσύνης κτλ. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δεν μπορούμε να εργαζόμαστε σε κοινωνία ε, εμπιστοσύνης όσο δεν έχουμε επιτάπητος θέση του όρους της εξειδίκευσης της πραγματογνωμοσύνης. Και χαίρομαι ιδιαίτερως κυρία Υπουργέ που εσείς κοινήσετε το ζήτημα της ε, αλήθειας, αλήθειας επιστημονικής ακρίβειας, αν και μπορεί το να βάζουμε στην ίδια φράση της λέξη επιστήμη και αλήθεια να γεννά πολλές φιλοσοφικές συζητήσεις. Ε, Πολλοί ήταν λοιπόν οι συνάδελφοι οι οποίοι ζήτησαν ε, ανα εξεταστική επιτροπή, ένα ζήτημα το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μας παρασύρει σε περίτες συζητήσεις. Πάνω απ' όλα πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είπε, τι είπε και γιατί. Γιατί την επόμενη φορά που θα έχουμε μια επιδημία και θα καλέσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί, δεν θα μπορούμε να τους πείσουμε γιατί ε, δεν θα έχουν εμπιστοσύνη πια σε αυτά που τους λέμε. Για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς επίσης, κύρια Πρόεδρε, θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας θέσεις, τις θέσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής βέβαια, ε, ε, σε σχέση με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, ως προς την επανεθνικοποίηση της ε, χρήσης των, των τροποποιημένων οργανισμών στην καλλιέργεια, γιατί εκεί πια είναι βέβαια γεωργικό ζήτημα. Όγκελεξ, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι έχουμε ακόμα ε, πολλά κοινά με τα οποία πρέπει να επιτελέσουμε τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και κυρία Γκροστέτ ε, ξέρω ότι έχετε εμπλακεί ε, στην έρευνα όσον αφορά την κινητικότητα των ασθενών την συνοριακή κινητικότητα και γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε δείξει ταυτόχρονα τη θέληση όλων των συναδέλφων ε, και, και, και εμού της ιδίας όσον αφορά το να γίνει ένα άνοιγμα και έτσι όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Και ταυτόχρονα, όπως ε, προείπα, ξέρετε ότι ότι εμείς έχουμε την βούληση να συνεχίσουμε την χρηματοδότηση ενός συστήματος παροχής τέτοιων υπηρεσιών και ο κύριος Ζιλ Μπαρνιό είπε ότι υπάρχει το θέμα του ιατρικού τουρισμού. Είναι πρόβλημα αυτό στη χώρα μας και σε ορισμένες περιφερειές της. Και πιστέψτε με, θέλω να αποσπάσω στο Συμβούλιο μια συμφωνία. Ήδη έχουμε αρχίσει τις επαφές. Προσωπικά έχω ασχοληθεί και θέλω να σημειωθεί συμφωνία. Και είπα προσοχή όσον αφορά την συστηματικοποίηση της προηγουμένης έγκρισης. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτοματοποίηση αυτή ε, σε μερικέ που υποχρεωτική, σε άλλε όχι. Γνωρίζετε ότι έχει ασχοληθεί με το θέμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Κοινοβούλιο στο παρελθόν επίση. όσον αφορά το να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο να μας προσφέρει διαφάνεια, ούτως ώστε να είναι δυνατόν να γίνει εκ μέρου των κρατών διαχείριση των θεμάτων τη υγεία και δεν θέλω να έχουμε αναδίπλωση όσον αφορά την συμφωνία του Ιουνίου. Δεν έχω πολλά περιθώρια λιγμού στο Συμβούλιο. Αυτό το ξέρω, το έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι, όμως θεωρώ ότι είναι ε, δυνατόν, είναι εφικτό και όσοι μιλήσατε το είπατε ότι θεωρείται δεδομένη μου την αποφασιστικότητα. Δρόσμα την παραποίηση των φαρμάκων θεωρώ ότι πρέπει να προωθηθεί το θέμα και οπωσδήποτε, εάν δεν κάνουμε τίποτα, εάν δεν κάνουμε τίποτα λέγω για την παραποίηση, ιδίω για να σταματήσουμε αυτά που γίνεται στο διαδίκτυο, τότε δεν προσέχουμε το διακύβευμα που είναι η υγεία των Ευρωπαίων. Άρα θέλουμε να κάνουμε τα πρόοδο και εσείς έχετε τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι χρειάζεται όπως λέτε στο ψηφισμά σας να έχουμε ένα άνοιγμα ε, να έχουμε μια πολιτική να προσέχουμε τι γίνεται στο διαδίκτυο Επομένως και σε αυτό το θέμα είμαι αποφασισμένη να προχωρήσουμε. όσον αφορά τις επαγγελματικές δεξιότητες έχουμε μια διάσκεψη ψηλού επίπεδου. Θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο. Θα μετάσχουν διάφορες επαγγελματικέ οργανώσεις. Θέλω να συνεργαστούμε και με τους ομολόγους μου πώς είναι με την απασχόληση γιατί εκεί είναι αυτό ο τομέας της λευκής όπως ονομάζεται εργασίας, όπου νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικέ προοπτικές και επομένω με αυτή τη συνάντηση υψηλού επίπεδου μπορούμε να διατυπώσουμε προτάσεις. Για το κάπνισμα. Οπότε δεν τελέστε θα γίνει μια τέτοια συνάντηση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να το παρατηθούμε. Και εγώ συμφωνώ 100% με τα όσα εσείς είπατε θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο να ενσωματώσουμε τις σχετικές προτεραιότητες ή στην ε, κοινωνική σχέση. Τώρα όσον αφορά τα φορολογικά μέτρα, ε, βεβαίως, και θα πρέπει να δούμε το, ότι υπάρχει εδώ πέρα ευρύτερη αρμοδιότητα όσον αφορά τη δημόσια υγεία, ε, αλλά τι να κάνουμε. Τώρα όσον αφορά το AIDS, Έχουμε τη διάσκεψη της επόμενης εβδομάδα στη Βιέννη. Εκεί πρόκειται να αναδειχθούν τα θέματα της ε, έγκαιρης πρόληψης. Τι ανάγκες υπάρχουν από φάρμακα. Sur Δεκεμβρίου είναι η παγκόσμια μέρα για το AIDS. Επίσης έχουμε και το ένα άτυπο συμβούλιο στο οποίο αναπτύσσεται μια Άλλη προβληματική, δεν ξέρω αν το έχετε και εδώ, είναι η, η αιμοδοσία. Ε, σε σχέση με τους ομοφιλοφίλους και με το AIDS. Οπότε θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτές τις διαφορές μεταξύ των Ευρωπαίων. να αποφύγουμε διακρίσεις διακρίσει κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά και θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χτενίζει ξανά το θέμα, να το συζητήσει από αυτήν την κρατημέλη, ώστε να δούμε πώ μπορεί να δημιουργήσουμε μια κοινή θέση. Για την γρήπη τα έναν ή ένα τώρα. Την πανδημία, όπω πολλοί είπατε. Θέλουμε να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια. ζήτησε εσωτερικό έλεγχο για το πώς έγινε η διαχείριση της κρίσης. Θέλουμε και εξωτερικό έλεγχο. Νομίζουμε ότι χρειάζεται μία πλήρης διαφάνεια. Έχουμε υποφέρει όσον αφορά την κατάτμιση των αρμοδιοτήτων αυτών που ασχολούνται με την κρίση και όταν ε, προέβηνε στις διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές βιομηχανίες είδαμε ότι υπήρξαν κάποιοι όροι, κάποιες ρήτρες που επευλήθησαν. Και αυτό γίνεται γιατί δεν διαπραγματευθήκαμε όλοι μαζί. Όχι, δεν γίνονται τα πράγματα έτσι όπως γίνεται σήμερα. Έχουμε πούμε δύο μέρες χώρες. Η μία ήθελε την, ε, τον εμβολιασμό μόνο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και άλλη ήθελε να γίνει αυτό σε όλους, ο εμβολιασμό σε όλους. Και δεν είναι ε, θέμα ε, επικουρικότητας, γιατί ας πούμε αν έχουμε μια πανδημία και ο όρος ακόμα είναι προβληματικός. Ξέρετε ότι τοποθετήθηκε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο άτυπο συνέδριο των Υπουργών στην άτυπη συνεδρία τους. Και όλοι, όλοι ας αναψάγουν στο Ιντερνετ τι γίνεται. Ε, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε με τέτοιο τρόπο την κρίση, τι γίνεται όσον αφορά την αποθήκευση των τροφίμων, τι γίνεται όσον αφορά τα εμβόλια, τι γίνεται τα, τα φάρμακα για τα ζώα, τι γίνεται για τα φάρμακα για τους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα επιμέρους, τα οποία βεβαίως εξελίχθηκαν. Άρα, θα πρέπει να δουλέψουμε με διαφάνεια. Ε, έγινε στις 2 Ιουλίου μια πρώτη διάσκεψη, εκπροσωπήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, υπέβαλε ερωτήσει προ, πρόεδρο του Κοινοβουλίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, το Συμβούλιο και είπε ο Επιτρόπος Νταλή ότι από τη μία μεριά έχουμε μια κοινή πλατφόρμα. Αυτό αφορά την ε, παραγγελία των ε, εμβολίων, αλλά από την άλλη μεριά είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια τέτοια διαχείριση που να είναι κοινή. Αφού όμως ε, συμπληρώσει την έκθεση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2011 και έτσι θα έχουμε τα συμβάσματα για όλα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες. Όσο και κυρία δεν θα πρέπει να ξεχνούμε όλα όσα έγιναν επί Ισπανικής Προεδρίας. Η Τρόικα, τι έκανα. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το πώς προχώρησαν τα πράγματα και η συνάδελφος ε, Ντοριέλ πρόκειται να σας ε, πει για κάποιες οδηγίες Όσον αφορά τώρα την ενημέρωση και την διαφήμιση, είμαι θέση να σας πω ότι όταν τα συζητήσαμε στο άτυπο συμβούλιο, το συζητήσαμε και κλεισμένον. τα μέλη του Συμβουλίου είναι ανοιχτά, επομένω υπάρχει ένα βήμα πρόοδο, θέλουμε να υπάρξει ρύθμιση, από μια μεριά της ενημέρωσης, από την άλλη της διαφήμισης, όμως σχεδόν όλα τα μέλη του Συμβουλίου είπαν προσοχή, μην έχουμε ως μασκαρεμένη ενημέρωση μια στην διαφήμιση. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε για να κάνουμε βήματα πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Υπουργό. Κύριε Λαγιέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Ρίσο. Η δυσκολία σε μια παρουσίαση είναι βέβαια ότι θέλοντας να είμαστε σύντομοι δεν μπορούμε να είμαστε και εξατλητικοί. Ναι, ευχαριστώ όμως για την ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία να απαντήσω. Νανοτεχνολογία λοιπόν είναι μια τεχνολογία. Ούτε καλή είναι, ούτε κακή. Πρέπει να την παρακολουθήσουμε, την αξιολογήσουμε και όταν χρησιμοποιείται σε τρόφιμα να εξασφαλίζουμε το ελάχιστο, δηλαδή την, την ασφάλεια των τροφίμων. Και γι' αυτό μαζί με τη Λάψκα και την Επιτροπή οργανώνουμε μια ειδική διάσκεψη για τις ανατεχνολογίες για τις 24 Νοεμβρίου που προφανώς είναι ε, προσκεκλημένα και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου τη επιτροπή αν το επιθυμείτε. Ε, νομοθεσία θα συζητήσουμε αν επαρκεί, εάν είναι εύστοχη, τις εφαρμογές της νομοτεχνολογίας και κάποιες από τις παρατηρήσεις σας ακριβώς αναφέροντας σε ζητήματα που έχουμε, προβλήματα που έχουμε και συμπεράσματα ως προς τις χρήσεις. Στις τρεις αυτές κατευθύνσεις λοιπόν θα προσπαθήσουμε τη διάσκεψη να δώσουμε απαντήσεις. Δεύτερον, όσον αφορά τους ε, ειδικού πραγματογνώμονες, σας μίλησα για τη διάσκεψη, είναι προφανές ότι ανεξαρτήτω του θέματος θα πρέπει να υπάρχει πνεύμα εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμοδίων λόγων τη αποφάση και των εμπειρογνώμονε. Και οι εμπειρογνώμονε θα πρέπει να έχουν και την ελευθερία να εκφραστούν, γιατί αν του χαλιναγωγήσουμε ε, και εκείνοι θα προστατευθούν πίσω από διάφορες, ε, διάφορα προσχήματα και δεν θα μιλήσουν ανοιχτά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ανοιχτά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα από το Βέλγιο για, τα, για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Έχουμε μια γνωμοδοτική επιτροπή για την χρήση και διάθεση στο εμπόριο των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η, η κυβέρνησή μας εμπιστεύεται αυτή την Επιτροπή Βιοασφάλειας και άρα μπορούμε να παρακολουθούμε τις εργασίες της και να τις ακούμε, να ακούμε τις συστάσεις της. Η ε, εμπιστοσύνη λοιπόν που θα πρέπει να εξασφαλιστεί ή και να ανακτηθεί σε ορισμένε περιπτώσει έχει τεράστια σημασία. Για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς Έχουμε σήμερα την έκθεση του κυρίου Ντάλι το απόγευμα. Ε, δεν μπορώ να σας πω λοιπόν πώς θα προκύψουν, πώς θα προχωρήσουν στο Συμβούλιο. Αλλά κάθε φορά που έχουμε να συζητήσουμε φάκελο ε, αδειοδότησης γραμματείων μικρών ε, στο Συμβούλιο Γεωργίας. Δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι η νομοθεσία που έχουμε είναι η πιο εύστοχη. και από την άλλη τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στη μειοψηφία, που θέλουν να καταψηφίσουν έναν τέτοιο οργανισμό και βρίσκονται στη μειοψηφία και αν εγκρίνει το οργανισμό, θεωρούν ότι τα παραγνωρίζουμε. Για την καλλιέργεια βεβαίω με πολύ μεγάλη προσοχή θα, προσοχή θα διαβάσουμε τι προτάσει του Επιτρόπου Νταλή που προτείνει την αρχή της επικουρικότητας. Εγώ προσωπικό γνώμη δεν έχω μένα, αλλά θέλαμε και στο, θα πρέπει και στο Βέλγιο να έχουμε μια άποψη και να αν δεν με ζήτημα των περιφερειών, αρμοδιότητας των περιφερειών στο Βέλγιο. Εν πάση περιπτώσει, ε, επικουρικότητα καλό θέλει είναι να μην υπάρχει, έστω και αν στην ουσία υπάρχει, στην πράξη υπάρχει. Η καλλιέργεια, παραδείγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν. Ε, επί παραδείγματι, αν δούμε στο Βέλγιο, στο νότο του Βελγίου ή στην Αυστρία ή σε άλλα κράτη ή περιφέρειες έχουν θεσπιστεί ε, νομοθετήματα τόσο αυστηρά που εκ των πραγμάτων απαγορεύεται η καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών, χωρί όμω ρητά να αναφέρεται αυτό και πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν έρθει να συζητήσουμε την αρχή τη επικούρικότητα. Έχουμε υπέρ μια όσο δυνατόν πιο ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, χωρί να η μετατραπεί αυτή σε μια κωδικοποίηση 27 ε, διαφορετικών εθνικών ε, νομοθεσιών. Νομίζω ότι ακόμα δεν βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ δεν είναι αρκετά ικανοποιητική η νομοθεσία στο βαθμό που είναι επικουρική αλλά δεν έχει το όνομα αυτό, έχει το τίτλο αυτό. κυρία Ντάκμαρ Ρότς Πέρεντ, σε δυόμιση λεπτά αν μπορείς να αρκεστείς Ντάκμαρ, κάν το τρία αν δεν μπορείς στα δυόμιση. Αδύνατο σχεδόν. Για το τομέα τη κυρία Όγκελινγκ στην υγεία καταρχάς, καταρχάς κυρία Όγκελινγκ, σας, ενημερώνω, σας ε, συγχαίρω για την ενημέρωση και το συνέδριο που οργανώνεται για το θέμα του Αλτσχάιμερ και την άνοια που είναι μια από τις μεγάλες απειλέ που αντιμετωπίζουν. Και για τα ε, παραποιημένα ή ε, παραχαραγμένα φάρμακα. Έχουμε πρόβλημα, όπως είπατε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, ε, ίντερνετ, πιστοποίηση, στοιχεία ασφάλειας. Στην ε, προσφορά υγειονομικής περίθαλψης χρειάζεται η ισοδύναμη προσφορά ασφαλειας στην προσφορα υγειονομικης περιθέλψης χρειαζεται περίθαλψης, το ίδιο και για την ενημέρωση του ασθενούς. Το θέμα που χαρακτηρίζει όμως την τοποθέτηση του Συμβουλίου, του Συμβουλίου είναι τα ε, οικονομικά, οικονομικές ανησυχίες. Τα κράτη-μέλη δηλαδή ανησυχούν ότι κάποιο μέτρο μπορεί να κοστίσει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα θέλανε. Αυτό το φοβίζει, όπως τα φοβίζει και στην... Ε, ε, υπερσυνοριακή παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και σε άλλα αντίστοιχα θέματα. Και ελπίζω, έχω σε εσά πολύ πολλές ελπίδες στηρίξη σε εσά ως Βελγική Προεδρία να ε, επαναφέρετε το αντικείμενο της συζήτηση στο συμφέρον του ανθρώπου, γιατί και ο άνθρωπος είναι κομμάτι της ιστορικής αγοράς. Ο άνθρωπος δηλαδή ο ασθενής και στην υγειονομική περίθαλψη όπως είπε και η κυρία Γκροστέτη, συμφωνώ ότι η πρόσβαση σε ισοδύναμη υγειονομική περίθαλψη είναι σημαντική πτυχή στην υπόθεση αυτή, αλλά τα κράτη-μέλη τα οποία δεν τολμούν να αγγίξουν το θέμα αυτό θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι μιλούμε για υγειονομική περίθαλψη ισοδύναμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν ε, πάρα πολλά πολύ διαφορετικές συνθήκες και προδιαγραφές ή πρότυπα πολλές φορές επέσχυντα ε, και άξια τρίτου κράτου, ε, του, τρίτου κόσμου στη, στα κράτη-μέλη και πρέπει να σημειώσω ότι ο πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου και αν ζει έχει δικαίωμα ένα, στην επιλογή του γιατρού του και στην επιλογή μιας ποιοτική υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό είναι που επιδιώκει το Κοινοβούλιο. Από την πρώτη μας ανάγνωση είπαμε ναι ότι πρέπει να υπάρχει το σύστημα της αδειοδότησης, η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να έχουν τον έλεγχο του σχεδιασμού τους κτλ. Τα είπαμε όλα αυτά και το δεχθήκαμε. Αλλά ταυτόχρονα ας μην ε, ε, φοβούμαστε μόνο τον οικονομικό Ε, ας μην φοβόμαστε μόνο το, το, τα, έξοδα, την οικονομική διάσταση. Ο κύριος Φέλνερ είναι εδώ, Συνάδελφο, τον είδα και νωρίτερα. Χαίρομαι που τον βλέπω εδώ, γιατί ασχολείται με τα θέματα αυτά και τα συμφέροντα των ασθενών, που πιστεύω ότι θα πρέπει πλέον να πέσουν οι εντάσεις και οι πιέσεις σε επίπεδο κρατών μελών και να μπορεί ο πολίτης πραγματικά να επιλέγει αυτή την υπηρεσία που θέλει. Ευχαριστώ κυρία Παρφάνοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτο ερώτημα για τις χρόνιες ασθένειες. Αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο θέμα στην παρουσίασή σας και στις προτεραιότητές σας. Ερώτηση θα εστιαστείτε επί συγκεκριμένων χρονίων ασθενειών και εκείνων που έχουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες και πέραν αυτού. Έχουμε 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες ε, που έχουν διάφορες μειοσκυλετικές ασθένειες. 49% προέρχονται, ε, οφείλονται άδειε ανάρρωσης σε αυτό. 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι απώλειες ε, για αναρωτικές άδειες, χαμένη παραγωγικότητα κλπ. Θα δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Όσον αφορά την ε, Ένωση για την Ψυχική Υγεία, κάτι, ένα θέμα πρόθεση Ισπανική Προεδρία. Θα το προωθήσετε κι εσείς. Δίνετε ιδιαίτερη σημασία στην αυτοκτονία. Στη Φλάνδρα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Merci. Peter Lise. Ευχαριστώ, Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω τρία σχόλια και εγώ να απευθύνω προς την κυρία Όγκελινγκς. Καταρχάς υποστηρίζω αυτά που είπε η Φρανσουάζο Γκροστέτ και η Ντάγμαρ Ροτ ε, Μπέρεντ για τα δικαιώματα των ασθενών και έχω κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα ήθελα να θίξω που εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε θετήσει τροπολογίες σχετικά με το θέμα. Όπου δεν, ε, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές επίπεδο συμβουλών και θα, προσπαθώ, θα παρακαλούσα την ε, κύριε Υπουργό να τα επαρεξετάσει τα θέματα αυτά. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε ορισμένες μορφές ασθένειες οι οποίες μπορεί να βρίσκουν λύση σε υπερσυνοριακό επίπεδο ή ιδεοντολογικές επιφυλάξεις. Δεν μπορούν να εκπλητερώνονται από την ε, δυνατότητα της υπερσυνοριακής ε, εξασφάλισης υπηρεσιών ή η προηγούμενη επιστοποίηση. Εάν όμως ε, ένας ασθενής κάνει τον κόπο να αισθήσει προκαταβολικά την ε, άδεια, δεν μπορεί να του ζητάμε να βάλει και το χέρι στην τσέπη επιπλέον. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να του δίνεται ένα πιστοποιητικό, ένα voucher ότι έχει κάνει ό,τι χρειάζεται και αναλαμβάνει το ταμείο του τα έξοδα. Να μην χρειάζεται δηλαδή να βάλει το χέρι στην τσέπη ο ίδιος. Στα ε, φάρμακα επίσης. Έγινε θέμα και με τις επανεισαγωγές. Στην ομάδα μου μας έχει απασχολήσει. Οι επανεισαγωγές λέμε δεν πρέπει να απαγορευθούν. Δεν τις θεωρούμε κύρια πηγή εισαγωγής παραποιημένων ή παραχαραγμένων φαρμάκων. Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την αγορά. Τώρα, γιατί είναι τόσο διαφορετική η κατάσταση στην αγορά των φαρμάκων μεταξύ κρατών μελών, γιατί έχουμε διαφορετικά μεγέθη, συσκευασίε, ε, μετρήσεις κτλ. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό σύστημα τυποποίηση. Μια ευρωπαϊκή αγορά των φαρμάκων μπορεί να μην μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσα σε ένα εξάμεινο, αλλά ίσως μπορούσαμε να δώσουμε το τριολάκτισμα Για δε την μόσχευση, μεταμόσχευση οργάνων πρέπει να συστήσουμε το θέμα αυτό που βέβαια έχει την ε, φαϊνή πλευρά του, δηλαδή την, ε, τη σωτηρία της ζωής ε, του ασθενούς, αλλά έχει και την φεά πλευρά του, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Ασία, όπου για λόγους, ε, και μάλιστα στην ε, Κίνα, όπου για λόγους μόνο και μόνο εξασφάλισης οργάνων προς μεταμόσχευση, γίνονται και φόνοι. Είχαμε τις, ε, την περίπτωση των εκτελέσεων μελών της αίρεσης Φαουν μόνο και μόνο για να χρησιμοποιηθούν τα οργανά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρία Στρέλλα. Εγώ έχω μία ερώτηση για την ε, Υπουργό κυρία Όγκελινγκ, την οποία και την ευχαριστώ για την εισηγησή της. Ε, θα ήθελα να επανέλθω αγαπητή κυρία ή στο θέμα που μας αναφέρατε, δηλαδή της κινητικότητας των ασθενών, ε, την διασυνοριακή κινητικότητα. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο το ότι εσείς ενδιαφέρεστε για το θέμα και ότι θέλετε να αποφύγουμε τον ε, ιατρικό τουρισμό. Όμως θα πρέπει και η επικουρικότητα να τηρηθεί και θα πρέπει επομένω να δούμε κατά πόσον μπορούμε να έχουμε μια σωστή χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων ε, και χρηματοδότηση σωστή. Και όπως ξέρετε έχουμε μεγάλες διαφορές από ένα κράτος στο άλλο. Αυτό αφορά την πολιτική για τα ε, συστήματα προνοίας. Αλλού υπάρχει, αλλού κοστίζει περισσότερο, λιγότερο, αλλού υπάρχει δωρεάν υγεία και είναι θέμα λοιπόν της κρατικής πολιτικής προγραμματισμού και χρηματοδότησης. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε και σε σχέση με το θέμα της προηγουμένης ε, έγκρισης πώς είναι δυνατόν να αλλάξουμε την κατάσταση, να έχουμε ε, μία προσέγγιση. Για κάποιε τέτοιε περιπτώσει θέλουμε να υπάρχει το σύστημα τη προηγούμενη έγκριση, ιδίω για, για κάποιες σπάνιες ασθένειες. Επομένως, ανησυχούμε για το πού μπορούμε να φτάσουμε όσον αφορά ε, κάποιες ε, διατάξεις που θα έρχονται σε σύγκρουση με κάποιες εθνική, εθνικές διατάξεις ε, που όμως προβλέπουν για κάποιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Τώρα, όσον αφορά κάποιες ε, ασθένειες που σχετίζονται με τις ασθένειες τη ρευματοπάθεια και σχετικά. Ε, εδώ μιλάμε για κάποια επίπτωση πάρα πολύ σοβαρή όσον αφορά την ε, οικονομία των κρατών μελών γιατί έχουμε δαπάνες άμεσες και έμεσε που προκύπτουν και πρόκειται για κάποιες ασθένειες που χτυπάνε τον κόσμο κάνουν τον κόσμο να μην μπορεί να, να, να κάνει τη, τη, δουλειά του σωστά αναγκάζει τον κόσμο να πάρει σύνταξη μια ώρα αρχίτερα με αυτές τις ρευματοειδείς ασθένειε. Βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση, αυτό θα βοηθούσε. Επίσης μια αγωγή ε, θα έπρεπε να, να, να βοηθήσει και να δούμε τι μπορεί να κάνει για τις, ε, τις σχετικές με τις ρεθμίες. Τι μπορεί να κάνει η Βελγική Πρόεδρια. Είπαμε ότι θέλουμε να υπάρχει μια πρωτοβουλία για αυτές τις ασθένειες. Άρα, ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Θα έχετε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ο επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι πρέπει να δώσω δίκιο στην ε, Dagmar Parents το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να έχει πάντα γνώμονα το οικονομικό κόστος και να περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής του, ασθενού ασθενούς ε, ή την ενημέρωσή του για τα φάρμακα που είναι διαθέσιμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ θα ήθελα για τα φάρμακα και για τη σχετική ενημέρωση να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Ξέρουμε ότι ήταν το πιο ακαθόδες θέμα αυτό και η αρχική πρόταση ε, δεν ήταν σύμφωνα με τις δικές μας προοπτικές. Θα θέλαμε λοιπόν μια επικοδομητική συνεργασία στο θέμα αυτό, μια κοινή θέση και ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή πρόταση να συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Ελπίζω με τη Βελγική Προεδρία να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά ώστε να έχουμε μια καλή λύση. Θα ήταν λυπηρό να αφήσουμε κατά μέρος το θέμα αυτό, να το αγνοήσουμε, να μην αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Ο Ευρωπαίος ασθενής χρειάζεται ενημέρωση. Καθημερινά την αναζητεί στο ίντερνετ. Αλλά είναι ενημέρωση από το ίντερνετ αυτή που βρίσκει, η οποία δεν είναι ελεγμένη δεν είναι πάντοτε ακριβής. Δεν έχουμε λοιπόν αρκετές πληροφορίες για τον ε, πολίτη. Και ελπίζω να γίνει συζήτηση επικοδομητική με το Συμβούλιο. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και εμείς και να ε, δούμε όλα τα θέματα Ελπίζω το Συμβούλιο να μην δώσει μόνο την εντύπωση ότι συζητά, Και ναι, μεν θέλουμε έναν καλύτερο ρόλο για τον ασθενή, σαφέστερο ρόλο για τον ασθενή, αλλά δεν μπορούμε να περιορίσουμε τα δικαιώματα του ασθενούς με μόνο γνώμονα το οικονομικό κέρδος ή όφελος. Ενημέρωση δεν σημαίνει πάντοτε μόνο διαφήμιση και εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ αν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε σε αυτή την, αυτές τις ρηπές των ερωτήσεων. Ομοφροντή ερωτήσεων μάλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω δεσμευτεί να κάνω τα πάντα για να πετύχω συμφωνία μαζί σας όσον αφορά τις υπερσυνεργικές αυτές υπηρεσίες που αποτελούν και αντικείμενο του ενθουσιασμού σας, της δουλειάς σας και της ε, βούλησής σας. Θα είναι εύκολο. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο όμως. Ναι, ξέρω πόσο ασχολείστε με το θέμα πόσο σας απασχολούν τα συμφέροντα των ασθενών, είναι σαφές ότι πρέπει να είναι η αφετηρία μας. Τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων ασθενών. Αυτό είναι προφανές κατά την άποψή μου. Αλλά αληθεύει ότι σε κάθε κράτος μέλος ξεκινάμε από διαφορετικά συστήματα υγείας. Πέρα από τα οικονομικά μέσα, τίθεται το θέμα της διαφοράς των συστημάτων. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Σε ένα λεπτό θα ήθελα να σα πω ότι γίνεται με το βελγικό σύστημα που ήδη το ξέρετε ίσω καλά. Ξέρετε ότι επενδύουμε πάρα πολύ όσον αφορά την περίθαλψη. Κάποιοι μα λένε συνεχώ ότι θα έπρεπε να επενδύουμε λιγότερα. Υπάρχει ετήσια αύξηση 4,5% αύξηση του προπολογισμού πέρα από τον πληθωρισμό για την περίθαλψη. Αυτό επί σειρά ετών. Βλέπετε για μας δεν κάνουμε οικονομίες πάση θυσία. Επενδύουμε σε προσβάσιμες ποιοτικές υπηρεσίες έχουμε ένα σύστημα πολύ ρυθμισμένο, πάρα πολύ ρυθμισμένο, προσβάσιμο τη πάση και σε ένα νοσοκομείο όποιος και να είναι η βασιλική οικογένεια είναι δίπλα στους άστεγους και έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα στον αφορά την περίθαλψη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και άλλα συστήματα είναι διαφορετικά και σίγουρα υπάρχουν και καλύτερα συστήματα από το βελγικό σύστημα. Ξεκινάμε λοιπόν πάντα από αυτές τις διαφορές. Προσπαθούμε να αποφύγουμε ε, τις ουρές που είναι προς, εις βάρος οι ουρές των ασθενών, εις βάρος των ε, δικαιωμάτων των ασθενών. Υπάρχει βούληση για την πράσινη των συμφερόντων του Ευρωπαίου ασθενούς. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε και ένα προστατευτισμό όμω οικονομικό. Θέλουμε να ακολουθήσουμε προσέγγιση που να υποστηρίζονται οι Ευρωπαίοι ασθενεί μη διαλύοντας ταυτόχρονα ένα σύστημα το οποίο θα ήταν εποφελές για τα συμφέροντα των Βέλγων ασθενών. Και νομίζω ότι όλοι μου οι συνάδελφοι με τον ίδιο τρόπο θα έλεγαν υπάρχει ένας τρόπος να πετύχουμε συμφωνία, είμαι πεπισμένη, ξέρω ότι θα είναι ευαίσθητο, θέμα κυρίως όσον αφορά το σύστημα των εκ των προτέρων αδειοδοτήσεων, τα ανέφεραν και άλλοι, ε, ε, α, της, πληρωμή πληρωμής κλπ, της προ, ε, προκαταβολής κλπ του κόστους. Όσο έχουν τα πράγματα. Τώρα που τον περασμένο Ιούνιο πετέφθη η πολιτική συμφωνία, είμαστε στις απάρχες, αλλά υπάρχει βούληση μαζί με το Κοινοβούλιο να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμφωνία που θα γίνει υπέρ των ασθενών. Αυτή είναι η βούληση που υπάρχει και επικρατεί. Όσον αφορά δεν έχουμε μια διάσκεψη όσον αφορά το θέμα της αυτοκτονίας. Είναι ευαίσθητη δύσκολη επιλογή. Σε κάποιες περιοχές της χώρας, ε, για κάποιες περιοχές ετοιμάζουμε ε, κάποια σχέδια πολύ φιλόδοξη να αντιμετωπιστεί αυτό. Υπάρχει μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου όσον αφορά τις χρόνιες ασθένειες από τη μια πλευρά και όσον αφορά ε, τις διάφορες ε, άγνωστες ασθένειες. Τι διαπιστώνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ότι όσον αφορά το θέμα αυτό είναι ξεκάθαρο ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ε, χρειάζεται πρόσβαση στην καινοτομία για τις ασθένειες αυτές, για τους ασθενείς αυτούς. Είναι σημαντικότατο πρόβλημα. Έχουμε εμείς ένα σύστημα αποζημιώσεως για τα φάρμακα, για το κόστος των φαρμάκων, αλλά πρέπει τουλάχιστον να ζητήσουν οι εταιρείε να υποβληθούν τα φάρμακα στη διαδικασία επιστροφή και γίνεται διαπραγμάτευση των τιμών. Και βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά ορφανά φάρμακα και οι εταιρείε δεν ζητάνε πλέον να μπουν στο σύστημα της ε, επιστροφής, της αποζημίωση. Όσον αφορά το θέμα αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βρούμε ένα σύστημα το οποίο θα πλαισιώνει αυτούς τους ασθενείς όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες ε, ξεκινώντας από αυτή τη διάσκεψη όσον αφορά τις άγνωστες ασθένειες και επίση και μια διάσκεψη όσον αφορά τις χρόνιες ασθένειες όχι αποκλειστικά διότι δύο βουλευτές είπαν προσοχή υπάρχει μια οικονομική πτυχή που σχετίζεται με την εργασία και την ε, παραμονή στην εργασία αυτών των ατόμων θέλουμε και λαμβάνοντα και αυτό υπόψη να ασχοληθούμε με την περίθαλψη και το κόστος της περίθαλψης των χρονίων ασθενούντων. Λοιπόν, και είπαμε όλα αυτά ξεκίνησαν τη διάσκεψη που θα γίνει αρχές ε, του φθινοπόρου. Όσον αφορά τις πληροφορίες, την ενημέρωση, με ρωτάτε αν έχω τη θέληση. Λέτε, βλέπουμε τις δυσκολίες όσον αφορά τους ορισμούς, ενημέρωση, διαφήμιση, ευθύνε που έχει η κυβέρνηση, η εξουσία, ε, ο ιδιωτικό τομέα κλπ. Και λέτε ότι ξέρουμε με βάση όλα αυτά τις παγίδες και τις δυσκολίες που πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή είναι και δική μου πεποίθηση. Όσον αφορά το θέμα αυτό έχω καθορίσει προτεραιότητες, καθόρισα προηγουμένως και πραγματικά και αυτό αποτελεί ένα κομμάτι από τις προτεραιότητες που έχω. Ιδού κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω σχεδόν για κάθε σημείο να σας πω και τι κάνουμε εντός Βελγίου. Και έχω καταλάβει τις τελευταίες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια υγεία ότι όσον αφορά το νομοθετικό πακέτο που αναφέραμε και που θίξατε ότι εκεί υπάρχει μια βούληση να κινηθούμε, να προχωρήσουμε σε συμπληρωματικότητα βεβαίως του εξαιρετικού έργου που έχει επιτελέσει αυτή η δική σας επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αυτά έχω να πω σε αυτά τις τοποθετήσεις σας. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για το ανοιχτό σας πνεύμα. Κυρία Λαγιουέλ, δεν υπάρχουν ερωτήσεις, οπότε ξαναπάμε Συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις. Η Σάρα Λότφορντ είναι ε, εκείνη που ξεκινά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ, λέει η Βαρόνι Λότφορντ ασχολούμαι με τις χρόνιες ε, ασθένειες, το θέμα το οποίο ανέφερε η συνάδελφος Παρνόβα. Και Έχουμε έναν φορέα για να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ε, διαβήτη, καρκίνο, ε, άλλες χρονίες ασθένειες και εγώ είμαι συμπρόεδρος αυτού του φορέα. Φυσικά και είναι διακομματικός. Χαίρομαι πολύ που θα ασχοληθεί με τις χρόνιες ασθένειες η Βελική Προεδρία. Έχετε προγραμματίσει τον Οκτώβριο επίσης αυτή τη ε, διάσκεψη, το συνέδριο. Βεβαίως ε, αυτό θα γίνει σε εβδομάδα Στρασβούργου. Και φαντάζομαι και εσείς θέλετε να ήμασταν εδώ, αλλά δεν θα είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε εδώ σε μια εβδομάδα συνόδου, άρα οι ευρωβουλευτέ δεν μπορούμε να πάμε στο συνέδριο που θα οργανώσετε. Πάντως, συγκεκριμένα θα ρωτήσω το εξή. Το Σεπτέμβριο του 2011 ο ΙΕ θα έχει μια συνάντηση υψηλού επίπεδου όσον αφορά τις ασθένειες οι οποίες ε, δεν είναι μεταδοτικές. Εμείς περάσαμε το Μάιο κάτι τέτοιο ε, σαν ψήφισμα εννοώ. Και υπάρχει και αυτή ε, η ειδική συνεδρίαση που κάναμε. Και τι γίνεται τώρα. Ο ΙΕ μάλλον θα ορίσει δύο μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων για να προετοιμάσουν εκείνη τη συνάντηση. Άρα θα έπρεπε να μετέχει η Ένωση με ένα από τα δύο αυτά κράτη-μέλη. Άρα εσείς τι ξέρετε σχετικά με αυτά. Γιατί θα πρέπει να συντονίσουμε τη δράση για να εκπροσωπηθούμε σε αυτήν την συνάντηση υψηλού επίπεδου. Γιατί θα έπρεπε να μετάσχει με ένα κράτος μέλος σε αυτή την κίνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Euh, Πρόεδρος, Σάρα, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Εγώ θέλω να αφαιρθώ στα ελάχιστα επίπεδα βοήθειας περίθαψης στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, καταλαβαίνω το κόστος, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες επίπεδα ελάχιστα βοήθειας. Βέβαια κάθε χώρα μπορεί να βελτιώσει αυτά τα ελάχιστα επίπεδα βάσει των δικών τους διαθεσιμοτήτων και των δικών του επιλογών κοινωνικών και υγείας όσον αφορά τα νέα τρόφιμα. Θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Ε, διότι στα θέματα που έθεσε στο, με τη χρήση των κλωνοποιημένου κρέατος και την ελεύθερη διάσταση στο εμπόρευμα και του κλωνοποιημένου κρέατος που προέρχεται από γόνους των κλωνοποιημένων ε, ζώων ε, ε, βρήκε αντίσταση στο Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σωστή η θέση όμως του Κοινοβουλίου πιστεύω. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δική σας θέση όσον αφορά αυτό το θέμα. Όσον αφορά τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την έκθεση που, που θα την έξω παρουσιάση Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το απόγευμα, διότι κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίζει ελεύθερα όσον αφορά τα προϊόντα, τα καλλιεργήσιμα στα εδάφη της. Ε, τουλάχιστον ε, γενετικά τροπένοι οργανισμοί που δημιουργούν πολύ προβληματισμό και ερωτηματικά. Όσον αφορά τη συνάδελφά σα για, μικρο... για την εργασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα ήθελα να ξέρω πώς προτίθεστε να προστατεύσετε την ευρωπαϊκή εργασία αυτό το εξάμεινο και να εγγυηθείτε στους νέους τη δυνατότητα να έχουν ένα μέλλον με εργασία εντός Ευρώπης και αν προτίθεστε να προχωρήσετε προς ένα δρόμο που θεωρώ σημαντικό, δηλαδή να ζητήσετε από τον, από από τον ΠΟΕ να ε, επιβάλλονται φόροι σε, τρίτες, σε προϊόντα που προέρχονται από τρίτε χώρε που δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων όπω στην Ευρώπη, διότι γίνεται έτσι αθέμητο ανταγωνισμό των επιχειρήσεών μου, άρα μπορούν να μειώσουν τι θέσει εργασία σε αυτέ τι αγωγέ και έναν φόρο άνθρακος πάντα α, επιπροϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό που δεν ε, καταπολεμούν ε, την αλλαγή του κλίματος, δεν συμμορφώνται με το πρωτόκολλο του Κιώτο, που είναι... Ε, δεν ασχολούνται τρίτε χώρε, επιχειρήσει των χωρών και δεν ασχολούνται με το περιβάλλον και άρα παράγουμε πολύ χαμηλό κόστο κάτω από το κόστο και εξάγουν τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνει παρέμβαση. Να επιβάλλονται φόροι στα σύνορα και θα ήθελα να ξέρω ε, ποια είναι η θέση σας όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Σέργιο Μπερλάτο. Και εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω μάλλον τις παρούσες υπουργούς και κλείνει το μικρόφωνο. Ε, με επιδεξιότητα παρουσίασαν το, τα προγράμματά τους. Το δικαίωμα στην υγεία των πολιτών ε, συνάδει και πάει χέρι με χέρι με το δικαίωμα της σωστής ενημέρωσης διότι πολύ συχνά η στρεβλή χρήση των πληροφοριών δημιουργεί περισσότερες ζημιές και από τους ιούς. Και από διάφορα επιχειρήματα ακούστηκαν στα, στις παρουσιάσεις και οι υπουργοί χρησιμοποίησαν μεγάλη σύνεση στη χρήση των λέξεων, διότι όταν μιλάμε για πανδημία της ε, νέας γρήπης H1N1, πανδημία είναι μια επιδημία μεγάλης κλίμακας. Και θα ήθελα να ρωτήσω τις δύο υπουργούς Ποια ήταν η επιδημία ευρεία κλίμακα που εξακριβώθηκε ότι υπήρξε στην Ευρώπη βάση επιστημονικών δεδομένων και όχι βάση λόγων. Και αν οι Υπουργοί έχουν στοιχεία όσον αφορά ε, τις ε, ανθρώπινων ζώων που αναφέρθηκαν ε, ε, που ε, οφειλότανε ε, στην ε, H1N1 e σε σχέση με τους θανάτους που αφιλόταν σε συνηθισμένη γρήπη. Όσον αφορά μετά τα εμβόλια, διότι ε, πρέ, αφορά την, την με, τα μεταβίβαση από άνθρωπο σε άνθρωπο προστατεύει αυτό το εμβόλιο της H1N1 Ποια είναι τα επιστημονικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Συμβούλιο Υπουργών που μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε με σιγουριά ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ε, το, ε, ο ιός του H1N1 και μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί προσεκτικότερα μια σίγουρη συνέπεια που είδαμε στην Ευρώπη με το θέμα H1N1 δηλαδή τον πολλαπλασιασμό τον λογαριασμών των εσόδων της φαρμακοβιομηχανίας που χρησιμοποιώντας λανθασμένη πληροφορία ε, ε, έβαλαν, απελευθέρωσαν διάφορα, διάφορους αντιγρυπικούς ιούς που δεν είχαν καμία σχέση με το νέο ιό της γρήπης. Όσον αφορά τον καρκίνο τώρα, όπως ξέρουμε η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και αυτό είναι σίγουρο και απόλυτο. Ρωτώ, ποιε είναι οι επενδύσει που προτίθεστε να κάνετε ώστε να εγγυηθείτε ότι θα δίδονται οι σωστέ πληροφορίε Δεν θέλω να αναφερθούμε τώρα σε πρωτοβουλίες κατά του καπνού, τέτοιους πρωτοβουλίες ή κατά του εινοπνεύματος ή κατά της ε, διατροφής, αλλά πρωτοβουλίες και επενδύσεις για να ενημερώνεται ο κόσμος όσον αφορά τις συνέπειες της κατάχρησης του καπνού ή των παραγόγων προϊόντων ή της κατάχρησης του εινοπνεύματος ή της κατάχρησης άλλων τροφίμων που λόγω της κατάχρησης αυτής προκαλούν μορφές καρκίνου που αν δεν εντοπιστούν εγκαίρως έχουν προφανώς ε, σε συνέπειες ανεπανόρθωτες. Θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα και από τις δύο υπουργούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπερλέτο. Η Άννα Ροσμπαχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ποια είναι η κατάσταση ως προς τη συνεχιζόμενη ε, αγωγή σε... Ε, ασθενείς. Ε, επίσης, στο ζήτημα των κλωνοποιημένων ζώων. Το Συμβούλιο. τι προσβλέπει, τι δυνατότητες δηλαδή για συμφωνία μπορεί να περιμένει όταν το Κοινοβούλιο έχει τόσο τι θέσεις. Για την ανατεχνολογία επίσης η οικονομική διάσταση φαίνεται να έχει προτεραιότητα έναντι τη υγείας μας και της ευημερίας είναι δυνατόν. Για δε τον καπνό και πέραν του καπνίσματος. Ο καπνός, ε, το ταμπάκο που λέμε, αυτό που βάζει κανείς στη μύτη για να, για να φτερνίζεται το σνους ε, που έχουμε στη Δανία, φαντάζομαι ότι ίσως είναι Ίσως, ίσως λοιπόν το σνούς αυτό να μην ε, ρηπαίνει το περιβάλλον, να μην ενοχλεί τους ε, άλλους, δεν εισπνέει κανείς άλλος ε, νοσηρά αέρια. Γιατί λοιπόν απαγορεύεται αυτό. Γιατί τους καταναλωτές θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ενημέρωση, αν υπάρχει σκοπός να ενημερωθεί ο καταναλωτής σωστά με κατάλληλα η σήμανση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ την κυρία Ρόσπαχ. Η Υπουργή Να αρχίσουμε την κυρία Λαριέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να σας πω όσον αφορά τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις συστάσεις Νταλή, με μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε τις ε, εργασίες του Κοινοβουλίου Οπότε στο Συμβούλιο θα ασχοληθούμε, θα το συζητήσουμε τέλος ε, Ιουλίου και να ζητούμε τώρα να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα συμβιβασμό. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για ελεύθερη κυκλοφορία ε, αγαθών, εμπορευμάτων, επομένως δεν είναι εδώ πέρα το θέμα μόνο η καλλιέργεια. Πρόκειται για για ελεύθερη κυκλοφορία να σας κάνει το κάθε μέλος, σας κάνει ό,τι της έρθει. Όχι, όχι, ε, θα πρέπει να το δούμε ευρύτερα. Τώρα γιατί για τους... Ε, για, το, για τις διαπραγματεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, υπάρχει εντολή διαπραγματευτική, έχουμε και διμερείς ε, επαφές και με τη Μερκοσούρ και επομένως κάθε φορά θα πρέπει να, να προσπαθούμε να δούμε ε, τι γίνεται κάθε φορά, ε, πού κερδίζουμε και πού χάνουμε ένα έδαφος και σε επίπεδο συμβουλίου. Προσπαθούμε να δούμε πώς όλη αυτή η προβληματική είναι δυνατόν σε επίπεδο ΠΟΕ να μας επιτρέπει να έχουμε με τέτοιες ε, διατάξεις που να μας βοηθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκό ε, να κάνουμε κάτι για τη δημοσία υγεία γιατί όλοι σήμερα θα πρέπει να καταβάλουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόστιμα προς τη ΣΥΠΑ γιατί υπήρξε αυτή η απαγόρευση όσον αφορά ε, τις ε, ορμόνες. Θα πρέπει όμως σε επίπεδο ΠΟΕ να γίνει αναγνώριση της ε, ιδιορυθμίας των ρυθμίσεών μας ότι θέλουμε ε, καλούν ταχύς των ζώων, έχουμε ε, κάποιες διατάξεις που επιβάλλουν το να, τηρούνται, να τηρεί την νομοθεσία για ό,τι εισάγουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Ευχαριστούμε κυρία ε, κυρία Υπουργέ, για αυτό που είπατε το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κυρία Όγκελινγκ, για τις άλλες ερωτήσεις. Όσον αφορά για το καπνό για μάσημα, σας παραπέμπω στην ερώτηση, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για αυτό που για την γρήπη. Είπαμε για αυτή την διάσκεψη του επίπεδου, η οποία μας έγινε και μας οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία συμπεράσματα αφορούν την εποπτεία, την επαγρύπνηση. Είναι αυτά στα οποία μπόρεσε να συμφωνήσει το Συμβούλιο και είπαμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτά τα κέντρα επιτήρησης ε, για την, σε επίπεδο επιδημιολογίας. Και όταν έχουμε κάποια κρίση να μπορούμε να έχουμε τόσα δεδομένα ούτω ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε χωρίς να πιέζονται πάρα πολύ αυτά τα κέντρα να δούμε τις επιπτώσεις της γρήπης και να δούμε τι γίνεται με τις πολυκλαδικές πτυχές του θέματος για να μπορούμε να μην έχουμε κενά στη γνώση μας, να ξέρουμε πού είμαστε ευάλωτοι. Να δούμε το πώς υπάρχει αλληλεξάρτηση των διαφόρων τομέων, κομματιών της κοινωνίας και της οικονομίας. γιατί είναι, θα πρέπει να έχουμε κάποια ανταλλαγή ποιοτικών πληροφοριών, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Άρα, να δούμε πώς με κάποιες προτάσεις, μέσα ακόμα και από άτυπες συναντήσεις κάτι θα καταφέρουμε και έτσι να δούμε τι ορισμοί θα δοθούν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Υγείας γιατί τονίστηκε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες των φαρμακοβιομηχανιών ανεξάρτητος όσον αφορά τα, τα, τα εμβόλια, όσον αφορά τις επιδημίες και να δούμε για τις κοινέ αγορές τι θα αποφασιστεί. Γιατί είδατε ότι αυτή η συνάντηση υψηλού επίπεδου έθεσε ένα αμφιβόλο το πώς δουλεύουμε, το πώς του τελευταίου μήνες προχωρούμε για να δούμε πώς η κάλυψη των εξόδων θα βελτιωθεί. Για τη συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά τον εμβολιασμό, είπαμε ότι η αρχή της οχροσύνης είναι το θεμέλιο της δουλειάς μας. Δεν θέλουμε να είμαστε με σταυρωμένα χέρια σε αυτή την ροή των πληροφοριών που επιταχύνονται σαν ρυθμός κάθε μέρα και ότι θα πρέπει επομένως να ετοιμαστούμε για το μέλλον, να θωρακιστούμε. Δεν είναι απλό Συνεχίσαμε με παθολόγους για τις ομάδες ψηλοκινδύνου και διαπιστώσαμε όσον αφορά τον εμβολιασμό ότι υπήρχε σημαντική πτώση θνησιμότητας όσον αφορά αυτούς που έπασχουν από εποχική ή εποχιακή γρήπη. Να, πώς προέκυψε ε, αυτό το αποτέλεσμα που αφορούσε την εποχιακή γρήπη. Πέραν αυτού τώρα, δεν είναι δυνατόν στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία εάν μας ξαναχτυπήσει. Βέβαια είπαμε παρένθεση αν θεωρήσουμε ότι έγινε πανδημία. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε το, το πώς δουλεύουμε, το πώς αντιμετωπίζουμε και επομένως θα πρέπει να αποκτήσουμε τα εργαλεία για να έχουμε διαφορετική μεθοδολογία πιάσαμε το αύριο κέρατα αυτή τη αρχή και είπαμε ότι κάνουμε 1η και 2η Ιουλίου αυτήν την διάσκεψη. 5 Ιουλίου το άτυπο συμβούλιο. Το βάλαμε στην ημερησία διάταξη. Επομένω, να, πώ ε, ασχολούμεθα εντατικά γιατί ξέρουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση. Τώρα, όσον αφορά τι χρόνιε ασθένειε. Και το ετώνησα προηγουμένω ότι όταν θα κάνουμε αυτή την προπαρασκευαστική διάσκεψη για όλες τις οσκελετικές ασθένειες στα πλαίσια της διάσκεψης για τις χρόνιες ασθένειες. Και γνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα παρουσίας και συμμετοχής των ευρωβουλευτών, μια ε, που έχετε τη σύνοδο στο Στρασβούργο, άρα να κάτσουμε να συνηθούμε να βρούμε μια άλλη ημερομηνία και να επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης και δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Στο άμεσο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά τον ε, καρκίνο είπαμε πολλά και μπορώ να σας πω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρονται πολλά για την πρόληψη γιατί είναι θέμα που καίει τους Ευρωπαίους. Θέλω να πάμε και στο επόμενο βήμα. Δηλαδή να υπάρξει και έρευνα. Το οποίο δεν έχει νόημα αν δεν υπάρξει αλληλεγγύη. Αυτό είναι προφανές. Και τελευταίο, όσον αφορά τις μη μεταδοτικές ασθένειες, είχα συμμετάσχει σε μια συνάντηση πριν από λίγους μήνες στην Γενέβη τον Φεβρουάριο για την πρώτη σύνοδο εκεί την πρώτη συνάντηση και ισχύει το ότι υπήρξε ευρωπαϊκό συντονισμό για να μπορέσουν αυτές τις πρωτοβουλίες να τις παρακολουθήσουν από κοντά γιατί παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά, κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος στον κατάλογο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Υπουργοί, για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Μπορούμε νομίζω να σας χειροκροτήσουμε όλοι. Πολύ καλή ποιότητα οι ανταλλαγέ απόψεων. Πολύ καλή ποιότητα οι απαντήσει και η ειλικρίνεια που είδαμε από πλευρά σα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν για μας το, ο τρόπος με τον οποίο η Βελγική Προεδρία σκοπεύει να αξιοποιήσει τους έξι μήνες της. Προτείνω να διακόψουμε για μερικά λεπτά, διότι θα έρθει ο Επίτροπος Δαλής στις 5. Yeah. καθίστε παρακαλώ. Euh, Υποδεχόμαστε σήμερα το απόγευμα με μεγάλη χαρά τον Επίτροπο Νταλή που θα μας μιλήσει για την πρόταση που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη και ανέκρινε όσον αφορά. Α, καταφθάνει ο Πρόεδρο, θα του δώσω το λόγο. Όσον αφορά την νομοθεσία για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann gerade da weitermachen. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζω. Από εκεί που σταμάτησε η κυρία Λεπάζ. Θα έρθουν αύριο από το Συμβούλιο η κυρία Σόφλιγκ να μας ενημερώσει για τις ε, εξελίξει το Συμβούλιο. Καλωσορίζω όμως εντωμεταξύ τον κύριο Νταλή, τον, τον Επιτρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ήρθε να μας ενημερώσει και με πολύ μεγάλη αδημονία περιμένουμε να ακούσουμε τι έχει αποφασίσει η Επιτροπή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, κύριε Νταλή. Σας δίνω λοιπόν το λόγο αμέσω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Αρχές του έτους, Μάρτιο του έτους 2010 ανέλαβε υποχρέωση να έρθω εδώ πριν το καλοκαίρι με συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με το πώς θα δώσουμε στα κάτι μέλη τη δυνατότητα να αποφασίσουν κατά πόσο θα επιτρέψουν καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην, στο εδαφό του. Χαίρομαι που έρχομαι να παρουσιάσω ένα πακέτο δέσμη μέτρων που εθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλι το πρωί και να το παρουσιάσω στην Επιτροπή σα στενή συνεργασία μεταξύ με εσά, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας εξασφ... αντικατοπτρίζουν σωστά τις ανάγκες και επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών. Οι προτάσεις είναι ένα, μια δέσμη μέτρων που επιτρέπουν δύο πράγματα, ταχεία και άμεση εφαρμογή λύσεων, που θα επιτρέπει αυτή την ελευθερία, την κριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη. Ασφάλεια δικαίου μακροπρόθεσμα ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν βάση επί της οποίας να κινηθούν ελεύθερα. Αυτή η νέα προσέγγιση όσον αφορά τους γενετικά του οργανισμούς, όπως παρουσίασα και πρόσφατα στους συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων, εφαρμόζεται μέσω των κάτω θυμέτρων. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, εξηγεί την πλέον ευέλικτη ε, προσέγγιση και προσέγγιση συνύπαρξης που θα αντικαθιστά την σύσταση 2003 από τώρα. Πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας 2001-18 την οδηγία περί καλλιεργιών όπως αποκαλείται για τη δυνατότητα που θα έχουν τα κράτη-μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τοπημένων οργανισμών στην επικράτειά τους κάτι που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου και πώς ερμηνεύεται αυτό ο πρόεδρος Μπαρόσο κατευθυντήριε γραμμές τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στο θέμα. Και είχαμε και έτοιμα κρατών μελών, 13 κρατών μελών, στο Συμβούλιο Περιβάλλοντο του Ιουνίου του 2009 να συνδυαστεί η αδειοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με το σύστημα με επιστημονική βάση με τη δυνατότητα των κρατών μελών να αποφασίσουν κατά πόσο θέλουν να καλλιεργήσουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμού βάσει άλλων λόγων πέραν των επιστημονικών. Το πρώτο άμεσο μέτρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα κράτη-μέλη χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία, ούτω ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τοπική, η περιφερειακή και η εθνική ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα μέτρα συνύπαρξη. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη νέα σύσταση περί συνύπαρξη. Ε, η πρότασή μα προβλέπει μεγάλη ευελιξία και αναγνωρίζει ότι τα μέτρα συνυπάρξεως που θεσπίστηκαν από τα κράτη-μέλη μπορούν α να έχουν σαν στόχο να έχουν χαμηλότερο κατόφλιο από αυτό που αποφασίστηκε τώρα στο 0,9%. Τα εθνικά μέτρα θα πρέπει να είναι ανάλογα με τον επιθυμητό στόχο, δηλαδή την προστασία των ιδιαίτερων αναγκών συμβατικών και βιολογικών καλλιεργητών σε κάποιες περιοχές και χώρες. Σαν δεύτερο βήμα το να δίνεται πραγματική ελευθερία στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν επί τη καλλιεργία των γενικά τροπημένων οργανισμών συνεπάγεται νομοθετική αλλαγή. Αυτή, αυτός είναι ο ασφαλέστερος νομικός τρόπος, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν λόγο όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικά τροπημένων οργανισμών με βάση πέραν της επιστημονικής αξιολογήσεως του περιβαλλοντικού και του κινδύνου για την υγεία. Τώρα, στην οδηγία για καλλιέργεια ένα συγκεκριμένο άρθρο για του γενικά του οργανισμού θα πετύχει το στόχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε αυτή τη δέσμη μέτρων με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Καλύψ, συναντηθήκαμε με όλου του ενδιαφερόμενου κατά την προπαρασκευαστική φάση και μέλη του Κοινοβουλίου και αντιπροσωπεί των κρατών μελών συναντήσαμε και αυτή η νέα πολιτική για την καλλιέργεια των γενετικά τροπημένων οργανισμών γενετικά του ε, έτυχε μέχρι τώρα θετικών αντιδράσεων. Αλλά όπως κάθε σημαντική αλλαγή ε, δημιουργήθηκαν και κάποια ερωτηματικά. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι έχω κάθε πρόθεση να συνεχίσω τις προσπάθειές μου για να βελτιώσω το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ενώση που βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία για γενετικά τροπημένου οργανισμού. Αυτό συμπεριλαμβάνει δράσει που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση τη αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων και τι απαιτήσει που έχουμε για τον έλεγχο των εγκεκριμένων σοδιών και καλλιεργιών. Θα δημοσιεύουμε την έκθεσή μας για κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες το τελευταίο τρίμηνο του 2010, κάτι που ζητήθηκε από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος το έτος 2008. Και συνεχίσουμε τις αξιολογήσεις οδηγίας περί καλλιεργιών και τον κανονισμό για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Επίσης, ε, έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε όσον αφορά τη φορολογική της οδηγίας άρθρα 26α και το νέο 26β όσον αφορά την υποβολή αναφορών και θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα που θα δοθεί. Καμία επιτάχυνση, καμία αποδυνάμωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας που συμφώνησαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το 2003. Συγκεκριμένες βελτιώσεις στη δύσκολη διαδικασία λήψεων αποφάσεων είναι κάτι που χρειάζεται κατεπηγόντως. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστούν τόσο ώστε να γεφυρώσουν τις αντίθετες απόψεις. Η νέα προσέγγιση όσον αφορά την καλλιέργεια γενετικά του ευθυγραμμίζεται με την πραγματικότητα και την πραγματικότητα των κρατών μελών. Και βάση της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας ακολουθούμε την προσέγγιση. Η λύση επιτάπητος αντιπροσωπεύει μια ισορροπία μεταξύ ε, αλληλεγγύης και μάλλον επικουρικότητας και του νέου πλαισίου που θέλουμε. Η νέα προσέγγιση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρωί είναι σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας έδωσα μια επισκόπηση ε, των βασικών ε, ζητημάτων. Τώρα προσβλέπω στο να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας και θα ήθελα να δώσω το λόγο, ε, να δώσω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον πρόεδρο της Επιτροπής σας. Τις προτάσεις που υθετήθηκαν σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Τζοντάλη για την ενημέρωση. επισκεφθήκαμε στην Πάρμα για μια αντιπροσωπεία την υπηρεσία. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα βεβαίως έχουμε. Ιδιαίτερος για την κατάρτιση των επιστημονικών μελετών, τις αναλύσεις, ιδιαίτερα για τον περιβαλλοντικό κίνδυνο ή κίνδυνο δημόσιας υγείας. Είπατε ότι υπάρχει ευρύτερη συνένεση, αλλά γεννούνται και αρκετά ερωτηματικά Νομίζω ότι σίγουρα τώρα θα ακούσουμε αρκετές ερωτήσεις. Είναι πολλοί οι συνάδελφοι που έχουν στήσει το λόγο. Ο κύριος δεν παραλαμβάνει να ρίξει πρώτος στο πυρ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον κύριο Νταλή που ήρθε να μας ενημερώσει όπως μας είχε υποσχεθεί πριν από ένα χρόνο. Ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχουμε την ε, ευκαιρία, πράγματι χάρη στη νέα νομοθεσία, να πιέσουμε και προς τα κράτη ε, μέλη και προς την Επιτροπή σε σχέση με τα θέματα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η συνύπαρξη λοιπόν ε, είναι ένας λόγος για τον οποίο απαγορεύεται η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Υπάρχουν στις προτάσεις της Επιτροπής κάποιες συγκεκριμένε ιδέες, ε, στις οποίες όμως θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες, εξηγήσει στη δικασία όπως έχει τώρα λοιπόν, γιατί μας είπε ο Επίτροπος ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν οι ε, διατυπώσεις ή οι διαδικασίες. Δεν πρόκειται δηλαδή να υπάρχει πιο χαλαρή διαδικασία για την ε, η επιτάχυνση της διαδικασίας για την αδειοδότηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Εδώ θα ήθελα πιο πολλές λεπτομέρειες και επίσης για το monitoring, την παρακολούθηση και τη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να λάβει περαιτέρω δράση για να παρακολουθεί με το monitoring τα φυτά τα οποία έχουν λάβει άδεια καλλιεργίας. Και επίσης στο μέλλον θα υπάρχει η ενημέρωση και η δυνατότητα για τον πολίτη και τι εμπλεκόμενε, ενδιαφερόμενες περιβαλλοντικέ ενδεχομένω οργανώσεις να παρακολουθούν την κατάσταση. Επίσης, στο κείμενο του Επιτρόπου υπάρχει ο όρος proportionate measures, αναλογικά μέτρα. Τι εννοεί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μιλάει για αναλογικά μέτρα στην περίπτωση της συνύπαρξης. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα, πρόκειται μήπως για μια συγκεκαλυμμένη ρήτρα που θα επέτρεπε ε, την, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να δώσουν άδειε για ορισμένε επιχειρήσει και, και γενετικά τροπημένου οργανισμού. Ευχαριστώ, κυρία Ροτμπέρεντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, ιδιαίτερα που ήρθατε να μας δώσετε την είδηση ακριβώ την ημέρα που ελήφθη η απόφαση Επιτροπή. Μερικέ παρατηρήσεις καταρχά. Σωστά λέτε ότι είναι προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα η νέα πρόταση. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα διοδότησης και τα κράτη-μέλη Υπάρχει διαδικασία διοδότηση και τα κράτη-μέλη μπορούν να απαγορεύσουν ε, ή να δώσουν ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν από την διοδότηση. Αυτό που λέγαμε μορατόριο παλιά, απλώ δεν είναι πραγματικά μορατόριου. Εν πάση περιπτώσει όμω, έχουμε την κοινωνικο-οικονομική αποδοχή σε ορισμένου κλάδου από την κοινή γνώμη και σε ορισμένου όχι. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι είναι αρκετά λογική. Σε ορισμένους τομείς όμως θα ήταν καλό να την συγκεκριμενοποιήσουμε, όπως πρότεινε μόλις ο κύριος Σέμπαχ για ένα τομέα. Η ε, ευρωπαϊκή αδειοδότηση, η αδειοδότηση μας λέτε, το σύστημα αδειοδότησης χρειάζεται βελτίωση. Μα προφανώς και εγώ θα συμφωνήσω. Είπε και ο πρόεδρος ότι επισκεφθήκαμε την ε, υπηρεσία, αποκεντρωμένη υπηρεσία τροφίμων και ασφάλειας ε, στην Πάρμα δεν αρκούν οι διατυπώσεις για την αδειοδόση αυτή τη στιγμή. Η αρχή της πρόληψης έχει ακόμη μπροστά της πολύ δρόμο και η κυρία Λεπάζη το γνωρίζει επίσης σε σχέση με την Εύσα δηλαδή βλέπουμε απαρέγκλητη ανάγκη για βελτίωση των ε, διαδικασιών και των αποτελεσμάτων. Δεν είναι αρκετά καλά αυτό αυτά που κάνουν στην ΕΦΣΑ, δεν έχουν κέρδη στην εμπιστοσύνη μας. Εσείς ήσασταν κάπως πιο διπλωματικός κύριε Επίτροπε βεβαίω και πρέπει να είσαστε διπλωμάτης εσείς, αλλά εγώ μπορεί να είμαι πιο ομή διότι αυτό περιμένει και από μένα πολύ τη τελευταία ανάλυση. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα διοδότησης καθαρό, δεν μπορώ να το πω βέβαια επικουρικότητα, απλώς θα έλεγα τα κράτη-μέλη μπορούν να λάβουν την απόφαση που θέλει ο πολίτης τους. Αλλά από την άλλη μετά έχετε δύο πυλώνες που κλείνουν το σύστημα. Καταρχάς έχετε το σύστημα περί νομοθεσίας ε, για την καλλιέργεια. Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχει και πρέπει να υπάρχει το σύστημα για την συνύπαρξη που αναφέρει και ο κύριο Σέμπαχ. Και είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες για την συνύπαρξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να υπάρχει η αδειοδότηση να υπάρχει αδειοδότηση την οποία μπορεί κανείς να ε, θεωρήσει ασφαλή, να υπάρχει δυνατότητα αυτή η λεγόμενη επικουρικότητα για τα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν την άδεια και στη συνέχεια να υπάρχει η κρίση σχετική με τη συνύπαρξη για χώρες στις οποίες, οι οποίες μοιράζονται μια περιφέρεια όπως μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου, Αυστρίας και Γερμανίας, Ιταλίας και α, Αυστρίας λοιπά Να μπορούν να συνεννοηθούν όταν σε μια περιφέρεια υπάρχει ο κίνδυνος ε, να επεκταθούν τα γενετικά τροποποιημένα ε, παρά τη θέληση του ενός του άλλου κράτους. Η κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Επίτροπο που να μας μιλήσει σήμερα. Συμφωνώ με τα όσα είπε η Ντάκμαρ. Έτσι θα μπορούσαμε να μέλη να προβούν σχετικές επαγορεύσεις και τώρα από πλευράς νομικής πέστε μας θα μπορέσετε να προχωρήσετε κύριε Επίτροπε. Δεν έχω δει την τελευταία εκδοχή του κειμένου αλλά η απαγορευτή γίνεται ούτε για συνύπαρξη, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για λόγους δημόσιας υγείας, τότε τι νομική βάση θα έχετε. Οπότε έτσι πάμε σε πάρα πολύ βάλλωτη ρύθμιση. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ε, το, υπάρχει ασφαλή δικαίωμα για τα κρατημένα τα οποία θα συμπλέψουν αυτή την απόφαση. Κάτι άλλο τώρα. Ε, ανησυχούμε όσον αφορά τις καινούργιες καθεντήριες που πρόκειται να συνοδεύσουν τη νέα διαδικασία. Ε, ο πρόεδρος Λάινεν και η Ντάγμα Ροτ Μπέρεν αναφέρθηκαν σε αυτή την ε, ε, ενδιαφέρουσα επίσκεψη που κάνατε στην ΕΦΣΑ και έγινε επομένως αυτή η ειλικρινή συζήτηση Μας είπαν βάσει της πείρας τους τι, τι προβλέπουν για τους τρομές οργανισμούς την ψημονική ε, ουδετερότητα και θεωρώ θετικό κύριε Επίτροπε αυτό που είπατε για το ότι θα πρέπει να έχουμε αμερόληπτους αντικειμενικούς επιστήμονες και ότι συμφωνεί Διευθύντρια της ΕΦΣΑ. Άρα θα πρέπει επί τη βάση αυτής της εμπειρογνωμοσύνης να κινηθούμε να αγκαλιάσουμε την πρόταση του Δεκεμβρίου του 2008 του Συμβουλίου που ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Και όσον αφορά επίσης τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων να έχουμε μια πολυκλατική ε, ολοκληρωμένη ε, εμπειρογνωμοσύνη. Επίσης ακούσαμε να μιλάτε κύριε Επίτροπε και για το περιβάλλον και τη σχετική υπερογνωμοσύνη. Σήμερα όμως δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι για την υγεία. Και άρα θα πρέπει να δούμε πώς οι νέες καυθυντήριε θα σας οδηγήσουν στο να χτενίσετε κάπως την κατάσταση για τις μελέτες για την ανθρώπινη υγεία. Μιλάμε για ένα τρίμηνο δεν μπορείτε να εκτιμήσετε τις επιπτώσεις, ιδίως των χρονίων ασθενειών. Άρα είναι πολύ βαριά η ευθύνη και πάρα πολύ εξημών θέλουμε να προχωρήσει η έρευνα στον τους τροπημένους οργανισμούς. Αλλά δεν αφορά αυτό μόνο την ε, ανάπτυξη. Αφορά τις συνέπειες των γενικά τροπημένων οργανισμών εις υγεία και περιβάλλον. Για αυτό που είπατε σε σχέση και με την προηγούμενη έγκριση για την ε, χλωρίδα και είπατε και η ΕΦΣΑ ενδιαφέρεται για αυτό το προϊόν. Όμως της, η ίδια η διευθύντρια της ΕΦΣΑ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει ακόμα να παρακολουθήσουμε για την Φλωρίδα. Στις 2 Μαρτίου δόθηκε έγκριση για αυτή την ποικιλία. Σας είπα ακριβώς όπως τα είπε η διευθύντρια της ΕΦΣΑ. Επομένως, εσείς συνεχίζετε και δίνετε έγκριση παρά τις επιφυλάξεις της ΕΦΣΑ η οποία επιφυλάχθηκε. Επομένως θα πρέπει η απόφασή σας να αναθεωρηθεί ή τουλάχιστον την ξαναεξετάσετε επιγόντως. Ευχαριστώ. Επόμενος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Χάση. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε να συζητήσουμε και θα πρέπει να σας πω καταρχήν ότι αισθανόμαι απογοητευμένη. Και ένας από τους λόγους είναι ότι συζητήσατε κύριε Επίτροπε προεβδομάδων το ίδιο θέμα με τους συντονιστές της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τότε τα είπαμε όσον αφορά το τι είδους εδάφη, τι είδους χώρους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να καλλιεργήσουν τροποποιημένα. Υπήρχε η φήμη, είχε κυκλοφορήσει ότι δεν θα τους επιτρέπατε και πολλά και μετά ότι δεν θα βάζατε υγειονομικούς και άλλους περιορισμούς. Τώρα βλέπουμε τη σημερινή πρόταση όπου παραμένετε, όπου δεν θεωρείται ότι μπορεί να επικαλεστεί ένα κράτος μέλος λόγους υγείας και λοιπά και περιβάλλοντος για να περιορίσει ή απαγορεύσει κάποιες καλλιέργειες μεταλλαγμένων Άρα μιλάμε τώρα για ευελιξία ενώ αφήνεται απ' έξω βασικά επιχειρήματα ε, με τα οποία θα μπορούσε κάποιο κράτο μέλος να περιορίσει τα μεταλλαγμένα, τα Επίσης, ήδη από το 2008 οι Υπουργοί Περιβάλλοντος ζήτησαν καλύτερη αποτίμηση, εκτίμηση κινδύνου. Δύο χρόνια πέρασαν σχεδόν. Μακρόπνοες επιπτώσεις. Τι γίνεται με τα ζενιοκτώνα. Τι γίνεται με τα φυτά που αντέχουν στα ζενιοκτώνα. Τα άλλα φυτοφάρμακα. πώς συμβιώνουν αυτά τα φάρμακα, πώς είναι εδώ να συνεπάρχουν. Και ότι θα πρέπει και για τους ανεξαρτήτους ε, ερευνητές να υπάρχει διαθέσιμη μια τέτοια ε, δυνατότητα εκτίμηση κινδύνου και όχι μόνο για κάποιες μεγάλες εταιρείε. Επομένως, τι γίνεται με αυτή την εκτίμηση κινδύνων είχαν ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα το Υπουργείο Περιβάλλοντο εδώ και τόσο καιρό και εσείς τώρα προωθείτε κάποιο μέτρο το οποίο προϋποθέτει μια σειρά εγκρίσεων για την καλλιέργεια μεταλλαγμένων. Μαρίζα Ματίας. Μαρίζα Ματίας. Ε, Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, αλλά ήδη τα ανέφεραν οι προλαλήσαντε. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν κάποια ζητήματα. Μετακινούμαστε από μια κατάσταση σε μια άλλη. από πλήρη απαγόρευση σε κατάλογο προϊόντων που θα επιτρέπονται. Θα ρυθμίζονται κάποια προϊόντα που θα επιτρέπονται και δεν θα ισχύσει πλήρης απαγόρευση. Είναι καλό που είναι εδώ επίτροπος. Είναι κρίσιμη σημασία η παρουσία του εδώ. Τέλος πάντων, θα ήθελα να υπογραμμίσω θέματα τα οποία ήδη αναφέρθηκαν. Χρειαζόμαστε εγγυήσει. Εγγυήσει για τους πολίτες μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες εγγυήσει, αρκετές εγγυήσει. Αυτό είναι θεμελιώδου σημασία όμως. Δεν είναι επαρκής, ανέφεραν οι προλαλήσαντες για ποιο λόγο. Και η νομική βάση έχει σημασία να μπορούν τα κράτη-μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, να το επιθυμούν. Άρα η, η σωστή νομική βάση είναι σημαντική. Δεν προσέχθηκε ιδιαίτερα η δυναμία της νομικής βάσεως. Δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα ερώτημα έχω, ή μάλλον είναι ένα θέμα χρονισμού που θα ήθελα να, να τονίσω. Ποιο είναι αυτό. Γνωρίζουμε όλοι ότι γνωρίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, προ... θα αποφάσιζε. Ξέραμε ότι θα ετοιμαστεί ανακοίνωση. Ξέραμε ότι θα χρειαστεί νέος κανονισμός, νέα νομοθεσία στον τομέα για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τέτοια επιτάχυνση της διαδικασίας της αδειοδότησης περιμένουμε όλοι νέα νομοθεσία, νέο κανονισμό. Και οι λόγοι που προευλήθησαν μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βιασύνη δεν είναι ξεκάθαροι. Γιατί τόσο η βιασύνη. Θα πρέπει να πριτανεύσει εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξηγήσει λοιπόν για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η βιασύνη. Χρειαζόμαστε διευκρινήσεις όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους δημοσιεύτηκε τώρα η ανακοίνωση. Ευχαριστώ. Τελειώνει εδώ πρώτος γύρος. Από τους συντονιστές και ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να είμαι σύντομος, ταυτόχρονα απαντώντας και σε όλες τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις που ακούστηκαν. η διάχυση της διαδικασίας. Καταρχάς σας διαβεβαιώ ότι δεν θα υπάρξει διάχυση διαδικασίας και δεν θα ε, υπάρξουν αδειοδοτήσεις χωρίς λόγο ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η Επιτροπή, όπως είπα και δημόσια, και νομίζω ότι το επαναλαμβάνει και κάποια κράτη-μέλη. Χρειάζεται δηλαδή, απαιτείται, η Επιτροπή θα ενισχύσει τη διαδικασία για την αδειοδότηση και την εφαρμογή των κανόνων για την αδειοδότηση. Επεξεργαζόμαστε ένα αίτημα από το Συμβούλιο για να ενισχυθεί η, περιβαλ... η πτυχή της του περιβαλλοντικού και ε, κοινωνικού αντίκτυπου αυτής της αδειοδότησης. Υπάρχουν όντως κάποιες καθυστερήσεις για διάφορους λόγους, αλλά πλέον περιμένουμε μέχρι το τέλη του χρόνου οι εκθέσεις για την ενίσχυση του περιβάλλοντος από τη χρήση των γενετικά τροπημένων οργανισμών να είναι έτοιμες, όπως επίσης και η αξιολόγηση αντικτύπου στο περιβάλλον και στην στη κοινωνία κοινωνικός αντικτύπος. Επίσης, ξεργαζόμαστε δύο ανεξάρτητες μελέτες για τη διαδικασία αυτή για να έχουμε ολιστικά τη θεώρηση της ε, εξέλιξης αυτής της διαδικασίας που θα κοιτάξουμε με επικριτικό πνεύμα. Ε, στο το τέλος του 2011-2012 νομίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα και να αντλήσουμε από αυτά τα συμπεράσματα ενδεχομένω με αλλαγέ στη σύλληψη. Μια ευρύτερη συζήτηση λοιπόν ε, για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς που χρειάζεται γιατί πρέπει με στη συζήτηση να εισρεύσει λογική, ορθολογισμός. Σας καθησυχάζω λοιπόν δεν θέλουμε να κατακαιρματίσουμε με επιτάχυνση και τα λοιπά τη διαδικασία. Δεν υπάρχει ζήτημα επιτάχυνση τη διαδικασία αδειοδότηση, ούτε ότι τα κράτη-μέλη θα υπερψηφίζουν την αδειοδότηση. Όχι. Εδώ είμαστε γιατί υποσχεθήκαμε ότι θα το κάνουμε. Το Μάρτιο είχαμε προσχεθεί ότι πριν το καλοκαίρι θα υποβάλουμε προτάσεις. Εργαστήκαμε εντατικά και εγώ και οι υπηρεσίες μου και ήρθαμε για την πρόταση. Περιτέρω αναφορά επιτήρησης, παρακολούθησης, ε, προτείνουμε πάλι ταχύτατα αμέσως να ενισχύσουμε τις στοιχές παρακολούθησης ε, των ε, μη κυβερνητικών, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, γιατί γνωρίζουμε ότι η επιστήμη μπορεί να εμπλουτιστεί. Οι γνώσεις επιστημονικές μπορούν να ε, διευρυνθούν, να εμβαθυνθούν και να καταστούν πιο χρήσιμες για το μέλλον. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι με το σύστημα αυτό του monitoring Εάν κάτι πάει στραβά, μπορούμε αμέσως να το αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό θέλουμε το ταχύτερο δυνατό να τεθεί σε εφαρμογή. Να μην περιμένουμε δηλαδή περισσότερο. Το ταχύτερο δυνατό να προχωρήσουμε και στο επίπεδο των Υπουργών για την εφαρμογή του. Και εδώ ζητώ συγγνώμη που θίγω διάφορα ζητήματα, αλλά μπαίνουν στην ίδια γραμμή και η ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ έχει σημασία. Επιμένουμε να υπάρχει ανεξάρτητη αναθεώρηση από επιστήμονες που συμμετέχουν σε ομάδες μελέτης ε, και έρευνας της ΕΦΣΑ ώστε να είμαστε σίγουροι για την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Για την αναλογικότητα. Και επί τη ευκαιρία μπορώ να απαντήσω και στην κυρία Χάση επί βάση μπορούν τα κράτη-μέλη να επιλέξουν να απαγορεύσουν την ε, καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Εμείς λέμε ότι μπορούν με οποιαδήποτε βάση να λάβουν την απόφαση αυτή. Δεν τους ελέγχουμε. Αρκεί να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το τι πράττουν. Αναλογικότητα σημαίνει απλώς ότι πρέπει να δοθεί μια αιτιολόγηση. Δεν μπορώ να λέει δηλαδή ένα κράτο, απαγορεύω του γενετικά τροπημένου οργανισμού γιατί δεν του γουστάρω. Όχι. Μια αιτιολόγηση χρειάζεται. Δηλαδή να πει θέλω να προστατεύσω την ε, βιολογική καλλιέργεια που έχω. Τη βιολογική χειρουργία. Ή η κοινή μου γνώμη αντιδρά υπερβολικά. Τάσεται αναφανδόν κατά των γενετικά τροπημένων οργανισμών και ούτω καθεξής. Ακόμα και τέτοια ζητήματα, δηλαδή κοινωνικο-οικονομικά ε, αίτια είναι για μας θεμητοί λόγοι απαγόρευσης της καλλιέργειας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Γιατί δεν αναφέρουμε την δημόσια υγεία και τους περιβαλλοντικούς λόγους. Να σας πω απλούστατα ότι αυτή η διαδικασία ξεκινάει από τη στιγμή που υπάρχει αδειοδότηση. Η διαδικασία της αδειοδότησης ήδη έχει ε, περάσει από μια επιστημονική γνωμοδότηση παιδοεύσα ΕΦΣΑ που εξετάζει τα, τους περιβαλλοντικούς ε, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Δηλαδή η ΕΦΣΑ άδεια θα δώσει μόνο και μόνο όταν υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ε, επικαλεστεί επιστημονικά κριτήρια για την επιλογή να μην επιτρέψει την καλλιέργεια. Τώρα υπάρχει και η δυνατότητα κανείς να προσβάλλει την επιστημονική κρίση της ΕΦΣΑ για, για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και, τον, και, τον, ε, και τη δημόσια υγεία. Και αυτό υπάρχει ήδη. Τώρα αυτό προσφέρουμε στα κράτη-μέλη ως βάση απόρριψης της άδειας ή απαγόρευσης καλλιέργειας είναι λόγοι μη επιστημονικοί πλέον έχουν και τη δυνατότητα να προσβάλλουν την επιστημονική κρίση, αλλά και πέραν τη επιστημονική κρίση έχουν τη δυνατότητα απλώ και μόνο να υπαγορεύσουν. Για την ε, υπερσυνοριακή συνύπαρξη. Η διασυνοριακή καλύτερα. Η διασυνοριακή συνύπαρξη, τα μέτρα δηλαδή αυτά, ήδη περιλαμβάνονται στις ε, τωρινές κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχει δηλαδή υποχρέωση για ενημέρωση αμοιβαία μεταξύ των κρατών των όμορων κρατών. και μέτρα ανάληψης ευθύνη σε περίπτωση επιμόλυνσης. Όλα αυτά μέτρα υπάρχουν για τους υπερσυνοριακούς ελέγχους ε, της συνύπαρξης. Αυτά συνεχίζονται, δεν αντικαθίσταται, δεν καταργούνται. Η πραγματικότητα τώρα που το αντιμετωπίζουμε σήμερα επίσης είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε 7 κράτη-μέλη, αν δεν ε, με πατάει η μνήμη μου, 7 κράτη-μέλη που με μέτρα διαφύλαξης ε, έχουν επιλέξει έμεσα, με τα safeguard measures δηλαδή, ε, απαγορεύουν την καλλιέργεια. αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι καθιστούμε πιο σαφή, πιο ξεκάθαρη την κατάσταση, πιο ασφαλή για τον καθένα δηλαδή. Δίνουμε στα κράτη-μέλη την ικανότητα να πούνε όχι στην καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών. Όχι περισσότερους γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Τα κράτη-μέλη έχουν πιο πολύ από ό,τι πριν τη δυνατότητα τώρα να λένε όχι στους γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Αυτό κάνουμε με τις οδηγίες αυτές. Για δε τη νομική βάση, η πρότασή μας είναι να υπάρχει δυνατότητα με τη νομική βάση τα κράτη-μέλη να καλύπτονται σε περίπτωση επιλογής του opt-out, δηλαδή απαγόρευση καλλιέργειας. Αυτή είναι η συμβουλή τουλάχιστον και της νομικής υπηρεσίας στην υπόθεση αυτή. Περιβάλλον, δημόσια υγεία, δεν μειώνουμε στην υπόθεση αυτή την ε, επαγρύπνησή μας συνεχίζουμε την παρακολούθηση των επιπτώσεων. Για την πατάτα ανφλόρα δεν μπορώ να πω τίποτα για την παρατήρησή σας. Είναι άγνωστο αυτό που είπατε. Σε μένα δεν το είχα υπόψη μου. Να ενημερωθώ όμως και αν υπάρχει κάποια ουσία ε, σε αυτό που είπατε, αν αληθεύουν δηλαδή οι ισχυρισμοί σας, θα επανέλθω. Επίσης ε, για την κυρία Ματίας επανέλχομαι. Mm. Για την ε, σπουδή με την οποία προχωρούν οι αδειοδοτήσεις. Όχι, δεν έχουμε σπουδή, ούτε μία σπουδή. Απλώς προχωρούν οι αδειοδοτήσεις όπως πρέπει. Πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία. Του να η διαδικασία αυτή έχει και συγκεκριμένα στάδια. Κανείς δεν πιέσει να συντομεύουμε τις διαδικασίες, κανείς δεν πιέζει για πιο γρήγορη χορήγηση άδεια, απλώς βλέπουμε ότι δεν μπορούμε ε, επαόριστο να περιμένουμε προκειμένου να λάβουμε μια απόφαση κάτι να συμβεί. Ε, όχι, γιατί διαφορετικά μένουμε σε έναν αέναο κύκλο αναβολής και δεν μπορούμε ποτέ να πάρουμε αποφάσεις. Ε, πρέπει να λάβουμε αποφάσεις, υπάρχουν διαδικασίες, πρέπει να βελτιωθούν έχουν αρχίσει να λαμβάνονται δράσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών. Σας διαβεβαίω δε ότι μέχρι τα τέλη του έτους θα ξανάρθω να σας δω για να συζητήσουμε όλες τις δράσεις που συζητούμε και αναπτύσσουμε προκειμένου να βελτιώσουμε το σύστημα και θα το βελτιώσουμε μαζί σας. Διότι πιστεύω ότι το επίπεδο της εμπιστοσύνης πάνω απ' όλα πρέπει να στοχεύουμε στη διαδικασία αυτή. Δεν μπορούμε δηλαδή κάθε φορά που συζητείται το θέμα των γενετικά τροπημένων οργανισμών να, ξεκινούν, να ξεκινούμε εμφύλιο πόλεμο. Πρέπει να προχωρήσουμε με καινοτομία αλλά με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο στην καινοτομία αυτή. Mm. Κύριος Λάινον, ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά δεν αλλάζουν πολλά πράγματα με τις νέες οδηγίες. Έχουν δηλαδή διασφαλιστική, είχαν μάλλον μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη τη διασφαλιστική δικλίδα. Τώρα και σε εθνικό επίπεδο έχουν τη δυνατότητα να πούνε το όχι μετά από μια αδειοδότηση. Απλώς διευρύνεται το φάσμα των λόγων για τους οποίους μπορεί ένα, ένα κράτος όχι στην καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών. Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύουμε αυτά που μας είπατε. Κύριος Ντάλι, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι. Ντάλι, επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ρήτρα διασφάλισης ήταν κίνηση από πλευρά των κρατών μελών. Και αυτή την κίνηση όφιλε να την αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν δεν την δεχθούμε αυτή την κίνηση, τότε ή τα κρατη θα πρέπει να διαγράψουν ή θα πρέπει να προσφύγουν στο δικαστήριο. Και έτσι αυτό δεν έγινε, οπότε η απόφαση των κρατών μελών δεν θα βρει αντίθετη την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Άρα είναι ακόμα πιο σαφή τα πράγματα. Ευχαριστούμε για την ευκρίνηση. Κυρία Αγιούσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε γιατί ήρθατε ταχαίως να μας εξηγήσετε την πρόταση αυτή την πρόταση την οποία γίνεται. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θέλει να ανοίξει τα σχήρα τη και θέλει να είναι το μπαλάκι στο γήπεδο των κρατών μελών. Γιατί τελικά δεν είναι θέμα επιστημονικό, είναι θέμα κοινή γνώμη. Ε, έχω ακόμα κάποια σημεία που δεν έχω καταλάβει, κάποια πραγματάκια να μου εξηγήσετε. Για ένα κράτο μέλο μπορεί να παράσχει μονομερός έγκριση ε, σε σχέση με ε, κάποιο τροποποιημένο ή είναι δυνατόν το, η Κομισιόν το κράτος μέλος να πούνε όχι σε αυτό το κράτος μέλος που το ζήτησε. Τώρα κάτι για την ιστορική αγορά. Μιλούμε κάτι μόνο για καλλιέργεια. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί ή μπορεί να του αρνηθούν την καλλιέργεια εν, ενός ε, τροποποιημένου ή αυτό αφορά και τη θέση σε εμπορία. Μπορεί ένα κράτο μέλο το οποίο καλλιεργεί να, να πουλήσει σε κράτο μέλο που απαγορεύει την καλλιέργεια του τροποποιημένου. Έχουμε την κοινή γνώμη, η οποία άγεται και φέρεται από φορτισμένες συναισθηματικά καταστάσεις και από την άλλη μεριά έχουμε το θέμα το επιστημονικό, το θέμα της δημόσιας υγείας. Γιατί με το τελικά την ύφη την πληρώσουν οι καλλιεργητέ. Έχουμε 130 εκατομμύρια εκτάρια τα οποία ε, ε, χρησιμοποιήθηκαν για, για τροπημένους του κόσμο και όλα αυτά μπαίνουν εδώ. Και εμείς εδώ λέμε για την ινσουλίνη, για την μπύρα, για, για ε, αυτούς τους μικροοργανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για κάποια τέτοια προϊόντα, ε, με, με, με οργανισμούς, μικροοργανισμούς. Ε, για το, το είπαμε αυτό για, για το βάβακα, χάσαμε την γνωστικότητα και τώρα ε, χώρε τρίτες χώρες κάνουν αυτά που εμείς ε, και εμείς κάνουμε το αντίθετο. Ενώ αυτοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτό το λεπιδόπτερο. για την ανταγωνιστικότητα. Πολλές φορές είναι τόσο ψηλό το κόστος που κάποιο τρόπο δεν συμφέρει να καλλιεργηθεί στην Ευρώπη. Όμως σόγια και αραβόστος εισάγεται μαζικά από τρίτες χώρες όπου τα τρόπο επιμένα συμφέρει να καλλιεργηθούν. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Τι είμαστε εδώ, μια φυσαλίδα, ένα, ένα κάστρο. δεν είμαστε, γιατί μπάζει από παντού αυτή, η φυσαλίδα, αυτό το, το κάστρο. Έχει παντού κερκόπρωτες και άρα θα πρέπει κάτι να γίνει γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε στο πρόβλημα. Έχω δουλέψει στην επιστημονική έρευνα για τα γεωργικά πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει κάποια καλλιέργεια κάποιο τροπημένο από την ΕΦΣΑ και από άλλους ε, οργανισμούς. Αν μπορούν να μου τον βρείτε, εντάξει. Ό,τι και να λέει η ετικέτα για το καλαμπόκι βάζουμε σαλάτα είναι τροποποιημένο. Αν λοιπόν υπάρχει τεκμηρίωση δεν έχω πρόβλημα. Όμως αυτό που με βασανίζει είναι ότι τελικά για όλα αυτά την ύφη την πληρώνουν οι αγρότες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Νταλή που ήρθε για να μας δώσει όλες τις εξηγήσεις του. Θα αναφερθώ και σε αυτά που είπε και η κυρία Γιούζο και εγώ. Δίνουμε μεγαλύτερη ελευθερία επιλογή στα κράτη-μέλη. Ξανά εφαρμόζουμε επιτέλους την αρχή της επικουρικότητας. Αλλά διερωτώμε. όταν μιλάμε για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, θα πρέπει να εντάξουμε τη συζήτηση αυτή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, της γεωργίας, της ευρωπαϊκής. Και δεν μπορούμε έτσι να αγνοήσουμε τον αντίκτυπο που θα έχει μια τέτοια προσέγγιση στην ΚΑΠ. Ξέρουμε ότι κάποιοι είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι καλή αρχή αυτή το να αφήνουμε την επιλογή στα κάτι μέλη, μπορεί να συμφωνούμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί αυτή περιπτώσει βολεύεται. Δεν υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Αφήνει την ελευθερία στα κράτη-μέλη. Αλλά εκτίθεται σε ένα κίνδυνο. Να δημιουργηθεί ανισορροπία μεταξύ των χωρών. Λόγω του αντιχτύπου των αποφάσεων των κρατών αντιχτύπων στην ΚΑΠ, για την ΚΑΠ και στρέβλωση στον ανταγωνισμού. Κύριε Νταλή, κύριε Επίτροπε, πέστε μας. Τι σκέφτεστε για αυτό το κίνδυνο που έφυξα. Θεωρείτε ότι είναι κάτι σημαντικό, εγώ έτσι πιστεύω. Εν τη αυτή περιπτώσει, πώς μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Αν Ντελβού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είμαι ευτυχέστατη. Ισύχασα από αυτά που μας είπατε όσον αφορά τη μη επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αυτό με καθησυχάζει. Η αρχή της επανεθνικοποίησης με προβληματίζει. Πολιτική κατά, κατά επιθυμία, κατά βούληση που επιτρέπει την καλλιέργεια και εμπορευματοποίηση των γενετικά του οργανισμών σύμφωνα την επιλογή των 100 μελών. Συμφιλιώνεται με την ενιαία αγορά. Συμφιλιώνεται με μια κοινή αγροτική πολιτική. Ομολογώ ότι εγώ έχω μεγάλα ερωτηματικά εδώ. Κυρίως όσον αφορά τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που ανέφερε και η Φρανσουάζ Γκοστέτ. Είχαμε τη Βελγίδα Υπουργό Γεωργία προηγουμένω που αναφέρθηκε στι ενδεχόμενε πρακτικέ συνέπειε αυτού. Μεταφορέ, Φερρυπίν. Μεταφορά γενετικών τροποποιημένων οργανισμών από μια χώρα που επιτρέπει του οργανισμού αυτού σε μια χώρα που δεν το επιτρέπει. Τι συνέπειε μπορεί να έχει αυτό. Πρακτικέ. Ανησυχώ αρκετά όσον αφορά τις... στο τι θα βαρύνει του ώμου των καλλιεργητών. Ποιε είναι οι νέε εγγυήσει που μπορούμε να του δώσουμε. Που θα εξασφαλίζει τη μη επιμόλυνση από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση. Αναφερθήκατε σε αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνεπειών, αξιολόγηση που έκανε η ΕΦΣΑ. Πώς θα διατηρηθεί η βιοποικιλομορφία. Η ΕΦΣΑ δεν έχει δίκτυα αξιολόγησης, αυτό στα υπόψη. Και πέραν αυτού, η ΕΦΣΑ δεν έχει ό,τι αξιολόγηση της χρησιμότητας των γενετικά τροπημένων οργανισμών. Δεν το ζητάμε αυτό, το ομολογεί η διεύσα. για την καλλιέργεια και την αδειοδότηση στην αμπόρια και για να μπορεί η Ευρώπη να χειριστεί το θέμα και να αναλύσει τον κίνδυνο, χρειάζεται άλλη προσέγγιση. Η αρχή της πρόληψης θα πρέπει να επικρατεί. Και κάτι άλλο. Γιατί να μην έχουμε απλούστατα να αποφασίσουμε να επικυρώσουμε την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Δεκεμβρίου 2008. Εκεί τα κράτη-μέλη οθέτησαν με την πλειοψηφία την ενίσχυση της αξιολογήσεως των γενετικά τροπημένων φυτών πριν από τη χρήση, να υπάρχει ετικεταθεσία στους πόρους και αυτονομία κάποιων ε, ε, γεωγραφικών περιοχών όσον αφορά την καλλιέργεια αυτή. Θα ήταν απλούστερο αυτό θα μπορούσε να εφαρμαστεί στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά τα ερωτηματικά έχει κύριε Επίτροπο, και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άντελβο. Ο κύριος Τρεμόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντέλη, συμμερίζομαι όλες τις ανησυχίες που εκφράζονται και σας ερωτώ αμέσως. Πόσο δημοκρατική είναι μια διαδικασία η οποία αγνοεί τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών ή τουλάχιστον της πλειοψηφίας και που ανοίγει τον ασκό του αιώλου και κάνει την επιμόλυνση από GMOs ένα ορατό σενάριο. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι αυτή η συμφωνία που προτείνεται είναι πρωτοφανής από την άποψη ότι ζητάτε να συνηγορήσουν στη γρήγορη και χωρίς ενδελεχή ανάλυση ρίσκου την έγκριση νέων ποικιλιών γενετικά τροποποιημένων με αντάλλαγμα να μπορούν να απαγορεύσουν αυτές τις καλλιέργειες αλλά δεν προστατεύει ούτε τους παραδοσιακούς, ούτε τους βιολογικούς καλλιεργητές, ούτε και το περιβάλλον. Στην ίδια την ανάλυση ρίσκου που κάνατε ως Επιτροπή, ανακοινώσατε ότι οι προτάσεις σας είναι πολύ πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους καλλιεργητές που δεν χρησιμοποιούν GMOs. Βεβαίω, με την πρότασή σας δεν δίνεται ταυτόχρονα στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να απαγορεύσουν την καλλιέργεια των ε, GMOs στη βάση κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όπως είπατε και πριν. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να απαντήσετε ταυτόχρονα, πριν φύγετε από εδώ, σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν τη νομική βάση. Ποια μπορεί να είναι λοιπόν η νομική βάση και πόσο στέρεη μπορεί να είναι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων. Και επιπλέον, εσείς ως Επιτροπή θα προσφέρετε τη νομική στήριξη που χρειάζεται απέναντι στις ΗΠΑ και τα άλλα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου όταν θα προσφύγουν ενάντια σε κάποιες χώρες μεγάλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν στην απαγόρευση. Τα ερωτήματα είναι σαφή και θα ήθελα να τα απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας κύριε πίτροπε. Κύριε Επίτροπε. Στο τελευταίο ευρωμαροβρόμετρο το 2005 για, τις, ε, για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξεπερνάει η έγκριση το 50%. Το πολύ πολύ 27% είναι η αποδοχή. Δηλαδή ένας στους τέσσερις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιο κράτος εγκρίνει, δέχεται τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς και ενισχύουν τα κρατη Πλην όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε τέσσερις φορές να άρει τι απαγορεύσει σε έξι κράτη-μέλη το 2005, το 2006, το 2007, το 2009, το Μάρτιο τελευταία φορά. Επίσης, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος έλαβαν ομόφωνη απόφαση για ένα σύστημα υπεύθυνο και αυστερό Φαίνεται ότι εσείς όμως προσπαθείτε να κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Επιτρέπετε για λόγους διοντολογίας την ε, ε, απαγόρευση, δηλαδή εισάγεται την αρχή της υπεκειμενικότητας. Θέλετε δηλαδή ίσως ε, να επιβάλλετε ένα σύστημα στο οποίο δεν, δεν θα είναι επιστημονική η όρη με τους οποίους θα απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροπημένων οργανισμών, ανεξάρτητα και επιστημονικά δεδομένα, αλλά θα στηριζόμαστε μόνο στην ΕΦΣΑ για, την επιστημονική κρίση και από εκεί πέρα θα έχουμε δοντολογική κρίση για το αν θα έχουμε την απαγόρευση όχι. Και επίση, η συνάδελφος το πας νωρίτερα ότι η επιλογή για μια απαγόρευση από κράτο μέλο, μόνο από λόγου, μη επιστημονικός εν πάση περιπτώσει ε, εισάγει την έννοια τη αβεβαιότητας ε, ως προς το δίκαιο που ισχύει. Θα ήθελα να μου δώσετε απαντήσει, λοιπόν. Η Επιτροπή θέλει το όντι να αποφύγει τις ανεκράτες επιστημονικές μελέτες. Αυτός είναι ο στόχος σας. Αυτό νομίζω θα μας απασχολήσει όλους και τους πολίτες πάνω απ' όλα. Ο πολίτη σε αυτό το συμπέρασμα θα καταλήξει με βέβαιος. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ που ήρθατε. Αυτό που θέλω να πω προκαταβολικά ως παρατήρηση είναι ότι δυστυχώς ε, ναι μεν ήρθατε να μας μιλήσετε αμέσως αλλά έχουν ήδη διαρρεύσει τον τύπο πολλά από αυτά που είχατε να μας πείτε και τα έχουμε διαβάσει από εκεί. Θα ήταν καλό ότι ενημέρωση είχαμε, δεν είχαμε απευθεία από εσά. Για δε τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς αυτό που έχω να πω είναι συγχαρητήρια γιατί είναι Πολύ καλέ οι προσπάθειε σας και είναι ντροπή και όνειρο για τα κράτη-μέλη ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις για την αδειοδότηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που έχει κρίνει ω ασφαλής η ΕΦΣΑ παρά τι επανελειμμένες επαληθεύσει και ελέγχου. δεν μπορούν να δεχθούν την αδειοδότηση τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή και στο παρελθόν ε, υποχρεώθηκε να ε, παραιτηθεί από αυτή την προσπάθεια. Αυτό όμως που έχω να πω, καλές οι ιδέες σας και η πρόοδος που ακολουθείτε, η πορεία που ακολουθείτε, αλλά θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα από την ΕΦΣΑ και πιο προσεκτική επαλήθευση ε, ότι δεν υπάρχουν επιρροές ή προβλήματα ανεξαρτησίας της κρίσης της, σε επίπεδο των συνεργατών της. Θέλουμε να είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή αδειοδότησης η ΕΦΣΑ. Ε, και επειδή ακριβώς η ανεξαρτησία της ε, τέθη έναν αμφιβόλο τα τελευταία χρόνια από αρκετά κράτη-μέλη και λόγω της συμπεριφορά των κρατών μελών ε, ή της αδυναμίας τους να προχωρήσουν σε αδειοδοτήσει, πρέπει σε αυτό το στοιχείο της ανεξαρτησίας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κατά τα άλλα, συγχαρητήρια για την πρόοδο που επιτύχατε. Υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα μέχρι τώρα και ε, αμφιβολίες, ανασφάλεια, αβεβαιότητα ως προς προϊόντα τα οποία δεν ξέρουμε αν έχουν αδειοδοτηθεί ή όχι και αν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης ε, μη γενετικά τροπημένων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. από τη δεκαετία του 90 όπου είχαμε ξεκινήσει με το μεγάλο πακέτο για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και είχαμε την πρώτη συνδιαλλαγή θυμάμαι ε, την περίφημη οδηγία για την απελευθέρωση, την οποία θεωρώ πολύ καλή ιστορία και επιτυχία, αλλά που τώρα πια έχει έρθει η ώρα να τροποποιήσουμε, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να διατυπώσουμε τα ε, στεναρά εκείνα επιχειρήματα, τα οποία θα μας επιτρέψουν και σε ορισμένε περιπτώσεις να απαγορέσουν τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς και να τους αδειοδοτήσουμε. Ερωτώ λοιπόν για την οδηγία για την απελευθέρωση. Τι άποψη έχετε τώρα, δηλαδή ποια θα είναι η μοίρα της. Θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ιδιαίτερα ε, με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα διότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι για λόγους καθαρά και μόνο αδειο, ε, ε, ιδεολογικούς και χωρίς καμία επιστημονική ή άλλη λογική βάση τάσσονται αναφανδόν κατά των γενετικά τροπημένων οργανισμών και της ε, τεχνολογίας, της γενετικής τεχνολογίας και, εξέλ, και της εξέλιξης και γι' αυτό θα έπρεπε να έχουμε μια σοβαρή τοποθέτηση. Επίσης, ε, διερωτώ με αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να ενημερώσει την κοινή γνώμη, γιατί δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Πολλές φορές θα το πω κάπως προκλητικά αν μου επιτρέπετε, φερόμαστε στον πολίτη σαν να είναι ηλίθιος. Προσπαθούμε δηλαδή μόνο να τον τροφοδοτήσουμε με φόβους αδικαιολόγητους ή αν τον κρατούμε δέσμιο. Ε, αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη, με μια εκστρατεία ενημέρωσης για τη, γενετικά, γενετική μηχανική να το αντιμετωπίσει. Πολλές φορές εδώ στην Ευρώπη έχουμε μια υπεροπτική τοποθέτηση στη συζήτηση για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς δεδομένης και της δημογραφικής ανάπτυξης και των κλιματικών αλλαγών σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως στα κράτη του τρίτου κόσμου. Έχω επίσης να ρωτήσω το εξής. Οι ελαστικοί κανόνες για την οδηγία για την ε, απελευθέρωση που θέλουμε να εφαρμόζονται. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα οδηγήσουν σε μια ε, απαγόρευση των γενετικά τροπημένων οργανισμών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είπε και η κυρία Ιούσο σε σχέση με τις αγωγές. Εάν πει ένα κρατοσμένος δεν θέλει αγωγές. Τι γίνεται. Και η γεωργία είναι αναγκασμένη πλέον η γεωργία μας να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, γιατί το 80% των πρωτοεμινούχων ζωοτροφών μας είναι εισαγωγέ. και μάλιστα από τι ΗΠΑ Πολιτείες στη Λατινική Αμερική, γενετικά τροπημένων οργανισμών, ε, προϊόντων. Γιατί λοιπόν ε, αρνούμαστε να συζητήσουμε το θέμα αυτό ανοιχτά. Η στη τελευταία ανάλυση και κόστο μεγάλο έχει αυτό. Η αύξηση των τιμών στα τρόφιμα πώς την κρίνετε εσείς. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να γνωρίσουμε. Όλα αυτά είναι ένα σύνολο που πρέπει να εξετάσουμε από κοινό. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Έχω ακόμη δύο συναδέλφους στον κατάλογο. Πέτερλε και Μαγκίνες, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ενδιαφέρον άκουσα αυτά που υπόθηκαν. Στη συζήτηση ήθελα να ακούσω για ποιους λόγους υπάρχουν εκείνοι που είναι κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Εγώ είμαι υπέρ. Από πλευράς επιστημονικής. Χρειάζεται μια νομοθεσία διαφανής να εφαρμοστεί στον τομέα. Χαίρομαι που υπάρχει και δυνατότητα τα κράτη-μέλη να πούν όχι αν δεν το επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους οργανισμούς. Αν ένα άλλο κράτος μέλος δίπλα από ένα άλλο πει όχι, ε, δίπλα σε εκείνο που λέει έχει πει όχι υπάρχει ένα άλλο που λέει ναι, ποια είναι η συνέπεια. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε σφαιρική θεώρηση όσον αφορά το θέμα. Ολιστική. Δεν ξέρω τι λέει ο Επίτροπος γι' αυτό. Νομίζω ότι ίσως αναφέρθηκαν κάποια τμήματα του ε, προβλήματος και της λύσης. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τομείς που αναλύουν περισσότερο ως πολιτική. Εγώ είμαι υπέρ της αναλογικότητας. Εκείνος που θέλει περισσότερο τους γενετικά οτροπημένους οργανισμούς και εκείνοι που βλέπουν μεγαλύτερους κινδύνους στους οργανισμούς αυτούς θα πρέπει να βλέπουν ότι οι θέσεις τους ε, λαμβάνονται υπόψη και είναι σεβαστές στην λήψη αποφάσεων. Ερώτηση. Μέχρι ποιου βαθμού η επιστήμη μπορεί να καθορίσει όλες τις διαδράσεις που μπορεί να υπάρξουν στη φύση, τις αλληλεπιδράσεις, μέσω της επικονίασης ε, μέσω των μελισσών η Εύσα δεν έχει απάντηση σε κάποιες ερωτήσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι τονίσατε κύριε Επίτροπε μια πιο επιστημονική προσέγγιση, αξιολόγηση του κινδύνου. Εγώ θα ήθελα απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Όταν ξεκινάει η συζήτηση γνωρίζω ότι τελικά τα στοιχεία γίνονται επιχειρηματολογία. Δεν αναφέρονται κάποιες πτυχές, αλλά μόνο τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται σε μια συζήτηση αντικειμενική. Και εγώ θα ήθελα, όπως η κυρία Σόμερ, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει την γενικότερη εικόνα και τις προπτικές όσον αφορά την πώληση αυτών των προϊόντων, την χρήση των γενετικών κάτροποποιημένων οργανισμών. Πιστεύω ότι είναι το ζήτημα και θα πρέπει να είναι προσεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να φτάσει στην καρδιά του προβλήματος και να το λύσει. Πάμε, αλλά θα πρέπει να κλείσω τον κατάλογο των αγοριτών γιατί ο χρόνος τρέχει. Η κυρία Μαγκίνες είναι η επόμενη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη κύριε Επιτροπή που δεν ήρθα όταν αρχίσατε την ομιλία σας. Διάβασα όμως τις ε, έντυπες δηλώσεις. Ε, ξέρετε, έπρεπε να πάω να συναντήσω κάποιους νέους ε, γεωργούς, τους είπα για τα μεταλλαγμένα και αυτό το οποίο ε, ήλπιζα ήταν ότι θα μπορέσουμε να τα πούμε καλύτερα, καλύτερα με τα κράτη-μέλη για τις νέες τεχνολογίες και για τα μεταλλαγμένα, διότι πάρα πολλές φορές το θέμα είναι ότι οι ε, επιστήμονες, οι ερευνητές θα πρέπει ε, να δούμε τι θα κάνουν όταν αρχίσουν οι απαγορεύσεις. Θα πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα ποιε είναι οι συνέπειες. Στην Ιρλανδία, τη χώρα μου, η κυβέρνηση, που δεν είναι το δικό μου κόμμα, ε, ψήφισε αποχή στο Συμβουλίο. Όμως, στην Ιρλανδία εισάγουμε ένα σωρό σόγια μεταλλαγμένη σαν πρωτεΐνη. Είναι εγκεκριμένη, είναι ασφαλής και δεν υπάρχει σήμερα κάποια απαγόρευση και δεν θέλουμε να σκεφτούμε στο μέλλον θα υπάρξει κάποια γενική απαγόρευση και έτσι η τεχνολογία να μας ωφελήσει αλλά και το κλίμα ωφελείται. Άρα ελπίζουμε ότι θα συζητηθεί καλύτερα το θέμα και όσοι όπως και εγώ είναι ανοιχτοί είναι δυνατόν να το συζητήσουν χωρίς να πρέπει ουσιαστικά να τσακωθούν Α, βλέπω. Χασκογελάτε. Χαχανίζετε, αλλά έτσι είναι. Είναι, είναι δύσκολη η συζήτηση αυτή. Γιατί από τη μία είναι η φανατική υπέρ και η φανατική κατά να γίνει ανοιχτή η συζήτηση. Και όπως είπε κάποιος συνάδελφος, όχι φορτισμένο ιδεολογικά, αλλά ρεαλιστικά. Δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε εξελίξεις που όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει αγκαλιάσει λογική προσέγγιση. Και αυτό είπα στους νέους ε, Γιώργους. Να γυρίσουν, να τα συζητήσουν με ανοιχτό πνεύμα. Και όλα αυτά να πάνε και στην κοινωνία. Και ό,τι πει η κοινωνία. και αν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν την καινούργια τεχνολογία, υποστούν τι συνέπειε γιατί πάρα πολλοί εδώ σε αυτή την αίθουσα ε, προβληματίζονται για αλλαγή του κλίματο και για το περιβάλλον. Όμω, ίσω αυτή η τεχνολογία μπορεί να μα ε, βοηθήσει. Δεν λέω ότι είναι πανάκια ή ότι θα λύσει το πρόβλημα τη πείνα στον κόσμο, αλλά ίσω λύσει κάποια από τα προβλήματα που έχουμε. Γι' αυτό και εγώ χαιρετίζω αυτή την ιδέα και ζητάω να υπάρχει πιο ανοιχτό πνεύμα. Ευχαριστώ κύριο Λύση, ο τελευταίο Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ήμουνα αρχικά κάπως επιφυλακτικό, αλλά ορισμένε από τι παρατηρήσει των συναδέλφων ε, με οθούν να λάβω και εγώ το λόγο. Για την υφιστάμενη οδηγία λοιπόν που εγκρίναμε και στο Κοινοβούλιο. Εγώ δεν είμαι σώτης της ε, γενετικής μηχανικής Θέλω να είναι αυστηροί οι κανόνες, να, είναι ασφαλής η χρήση, η χρήση, αλλά πρέπει να πω ότι έχουμε τους πιο αυστηρούς κανόνες του κόσμου. Δεν υπάρχουν πιο αυστηρές συνθήκες αδειοδότησης στον κόσμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον και δεύτερον και πολιτική επιτήρηση, ε, παρατήρηση. Ποτέ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποτέ έκτοτε δεν είχαμε ε, τόσους πολλούς πράσινους υπουργούς στην, στο τραπέζι του Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος όσο τη στιγμή που λήφθη σχετική απόφαση για την οδηγία αυτή. Γαλλία, Ιταλία, ε, Σουηδία, Γερμανία και δεν ξέρω ποια άλλη χώρα ήταν όλοι οι υπουργοί από πράσινα κόμματα. Επομένως έχουμε τις καλύτερες εγγύησεις αυστηρότητας για τα κλωνοποιημένα. πρέπει το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τις αποφάσεις που λάβαμε, πρέπει να έχουμε λογικά επιχειρήματα και τα κράτη-μέλη τα οποία ε, διστάζουν στην περίπτωση των γενετικά τροπημένων οργανισμών ε, θα διστάζουν προς την αδειοδότηση. Δεν μπορεί βέβαια να τα υποχρεώσει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και παρακαλώ όλοι μαζί να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φύλακα των συνθήκων και των υφισταμένων νομοθεσιών και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι όταν κάποιος δεν έχει επιχειρήματα στεναρά, επιστημονικά βάσιμα για μια απαγόρευση, να τον προσαγάγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την αυθαιρεσία. Εάν ένα κράτος μέρος δηλαδή το οποίο δεν ε, δεν έχει σοβαρούς λόγους, απαγορεύει για πολιτικούς μονολόγους την ε, αδειοδότηση, θα πρέπει να το παραπέμπουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και όταν πια υπάρξει ε, μελέτη, επαρκής μελέτη και τεκμηρίωση ε, για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ναι, πρέπει να επιτρέπεται να χορηγείται η άδεια. Εάν ακολουθήσουμε τη μέθοδο που προτείνετε εσείς, θα έχουμε το εξή φαινόμενο, το προβλέπω, ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια επιχείρηση να κάνει την προσφυγή στο δικαστήριο στη θέση σας και τότε θα είναι ίσως πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, για άλλη μια σειρά, μια φορά, μια σειρά από παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το αντικείμενο που συζητούμε και η πρότασή σας. Ελπίζω η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι προς την επανεθνικοποίηση. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα λύνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη και για την ιστορική αγορά και για τη γεωργία και τη γεωργική αγορά και για τις όμορες περιφέρειες, το αναφέρατε εσείς νωρίτερα, τι συνέπειες θα έχει να προβλεφθεί η μη η αδειοδότηση και η χρήση αυτών των προϊόντων. Κάποιοι συνάδελφοι υπέκριναν την Εύσα. Μετά την επίσκεψή μας στην Πάρμα, εγώ υποχρεούμε να διαφοροποιηθώ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς το σε τι διατυπώνουμε επικρίσεις για την ΕΦΣΑ. Επιστημονικό Συμβούλιο 21 διακεκριμένων επιστημόνων, διαλεγμένων, ένας προς έναν διαλεγμένοι, με την ε, βέλτιστη κατάρτιση, με δεδηλωμένη ανεξαρτησία. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι δεν είναι, ότι δεν ανεξάρτηση, ανεξάρτητη. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε πιο επικριτικά το τι γίνεται με τις αναλύσεις της ΕΦΣΑ. Συνέπειες για τη δημόσια υγεία, όπως είπε και ο κύριος Πέτερλε, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον σε περίπτωση απελευθέρωσης. Υπάρχουν επαρκείς μελέτες για τις συνέπειες αυτές. Εκεί ίσως πρέπει να είμαστε πιο επικριτικοί. Αλλά πάντως προκαταβολικά δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν είναι ανεξάρτητη η ΕΦΣΑ. Δεν, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο ανεφετέρου. Μπορεί κάποιο αποτέλεσμα μελέτης να μην μας ικανοποιεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, έχει απολέσει την ανεξαρτησία της. Η κυρία Ζόμερ λέει ότι πρέπει να ενισχυθεί η αξιοπιστία ή η φήμη της ΕΦΣΑ και από την άλλη λέει ότι θα πρέπει να προσάγουμε τα κράτη όταν δεν ακολουθούν τις συστάσεις της ΕΦΣΑ. Ε, κάπου είσαστε... Είναι σόλικο αυτό που είπατε κυρία Ζόμερ, ο Επίτροπος. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τα πολλά σχόλια που ακούστηκαν. Άκουσα όλα τα σχόλια και θα πρέπει να τα αναλύσουμε και ελπίζουμε να είμαστε θέση να συζητήσουμε πολλά από τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το την ύπτη σχήρας της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ των ευθυνών που συνεπάγονται σε αποφάσεις πρέπει να πω ότι η ευθύνη είναι πράγματι η ευθύνη των κρατών μελών που, δεν, ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη ποτέ δεν ε, ε, ενέκριναν κάποια απόφαση περί των οργανισμών αυτών, ούτε και δεν ενέκριναν ή απέρριψαν απόφαση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πάντα τα κράτη-μέλη κατέληγαν σε μία απόφαση αφήνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λήψη της απόφασης. Άρα δεν τίθεται θέμα το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νύπτει τα σχήρας της, αλλά να αναλάβουν αυτοί που πρέπει τις ευθύνες τους. Και εδώ είμαστε ευαίσθητοι. Ευαίσθητοι λέγω κατανοούμε τις πραγματικότητες που επικρατούν σε διάφορα κράτη-μέλη και δεν μπορεί να είναι μία ενιαία λύση αυτή που θα χρησιμοποιηθεί. Αναφέρω τη χώρα μου, μία μικρή χώρα, 320 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο σύνολό της. Τι κανόνες μπορεί να θεσπίσει εκεί για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, για τη συνύπαρξη. Ένα παράδειγμα, άλλη χώρα, που προωθεί την αγιατική της οικονομία προς τη βιολογική καλλιέργεια, εκτατικά. Άρα θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις και δεν θα πρέπει να τις επιβάλλει άποψη η βιομηχανία που επιμένει να καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς εν το μέσο των βιολογικών καλλιεργείων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που λέμε είναι ας είμαστε λογικοί. Ας καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση. Δεν είναι θέμα επανεθνικοποίησης της αγοράς. Αλλά δίνουμε την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι θα συμβεί στην επικράτειά τους. Εδώ μιλάμε για καλλιέργεια. Είναι σαν να κατασκευάσει ένα κτίριο αν θέλω να πω θα φτιάξω ένα εμπορικό κέντρο και έχω εδώ το σχέδιο για ένα εμπορικό κέντρο και είναι πολύ καλό, αποτελεσματικό και θέλω να το οικοδομήσω όπου θέλω, δεν με τρέπεται, διότι κάθε κράτο μέλος μπορεί να μου πει αν μπορώ ή δεν μπορώ να κτίσω στην επικράτειά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε και σε πολλές άλλες περιστάσεις. Ας το δούμε έτσι. Δεν συζητάμε το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αυτό κάθε αυτό αλλά το δικαίωμα που δίνουμε στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να μην καλλιεργήσουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό τίθεται, αυτό προτείνεται σε αυτή τη φάση. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Για να απαντήσω στην κυρία Αγιούσο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθεί να, χωρί, να λαμβάνει τι αποφάσει αδειοδότηση για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, δεν θα υπάρχει αυτοεξαίρεση όσον αφορά το εμπόριο. Το εμπόριο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα είναι εντελώ ανοιχτό, θα είναι ελεύθερη αγορά. Οποιαδήποτε χώρα καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένου οργανισμού μπορεί να του πουλάει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. I agree with... Συμφωνώ μαζί σα και με την κυρία Γκροστέτ. Πράγματι, όπως είπατε, δεν μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη μια φυσαλίδα που προστατεύεται από την καινοτομία. Το τόνισα και το υπογράμμισα τους μήνες που είμαι σε αυτή τη θέση. Και το είπα και σε αυτή την επιτροπή. Δεν θα είμαι εγώ υπεύθυνο για να ρίξω την ε, Ευρώπη στα λιμνάζοντα νερά στον αφορά την καινοτομία. Αυτό θα ήταν αντίθετο προς τα συμφέροντα του Ευρωπαίου πολίτη. Πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία. Όμως θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που απορρένω τις πράξεις μας και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαδικασία αξιολογήσεως των ελόγω κινδύνων. Γι' αυτό στη, παροτρύνω στις παρεμβάσεις μου λέγοντας ότι θα πρέπει να έχουμε υπεύθυνη καινοτομία. Καινοτομία που όπως αναφέρθηκε θα μας λέει και ποια είναι τα ωφέλη για το πληθυσμό από την καινοτομία. Πρέπει το ξέρουμε αυτό, διότι η καινοτομία σαν αυτοσκοπός για το βραβείο Νόμπελ ή για κέρδη για μια εταιρεία δεν είναι καινοτομία που θα ήθελα εγώ. Θα ήθελα εγώ να δω καινοτομία που είναι πραγματικά επωφελής για την ανθρωπότητα εν γέννη, για τα ανθρώπινα όντα. Και υπάρχουν πολλές δυνατότητες στον τομέα που συζητούμε. Ακούσαμε και αυτά που μας είπε η κυρία Μακίνες ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό, αλλά θα πρέπει να δούμε πραγματικά ποιε είναι οι δυνατότητε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και να τα σταθμίσουμε. Δεν είμαι υπέρ κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ιδεολογικά δεν είμαι τοποθετημένο υπέρ μια πλευρά. Αλλά πιστεύω ότι έχω την ευθύνη να δω τι γίνεται μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμε, ποιε θα είναι οι συνέπειε ε, των αποφάσεων που λαμβάνουμε σήμερα. Όσον αφορά τη νομική αβεβαιότητα, την ασφάλεια δικαίου. Εγώ επέμεινα να ακολουθηθεί η διαδικασία συναπόφασης. Ακριβώς γι' αυτό. Για να τοποθετηθεί σωστή νομική βάση στα όσα κάνουμε. Για τις αποφάσεις που θα λάβουν τα κράτη-μέλη. Θα υπάρχει νομική βάση για αυτοεξαίρεση από πλευράς κρατών μελών. Και εγώ θα υποστηρίζω τα κράτη-μέλη και έναντι των ΙΠΑ και έναντι του ΠΟΕ, κράτη-μέλη που θα αντιταχθούν σε αυτή την προσέγγιση, διότι πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ίδιο πιστεύει, ότι είναι η σωστή προσέγγιση που ακολουθούμε. Με ρωτήσατε γιατί να επιτρέψουμε αυτοεξαίρεση που βασίζεται σε επιχειρήματα περιβαλλοντικού κινδύνου και υγείας. Το επανάλαβα αυτό. Ο πιβαντικό κίνδυνο και απειλή για την υγεία θα έχουν ξελογηθεί από την ΕΦΣΑ ήδη όταν χορηγείται μία άδεια. Αυτή η διαδικασία ξεκινά μετά την ε, αδειοδότηση, άρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτοεξαίρεση βάση θετική αποφάσεω για να πάμε αντίθετα στη θετική απόφαση τη ΕΦΣΑ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι λόγοι βάσει των οποίων θέλουν αυτοεξαίρεση τα κράτη-μέλη. Αν θέλουν να επιμείνουν για λόγου υγεία και για λόγου περιβάλλοντο αυτοεξαίρεση, opt-out, τότε εξακολουθούν να έχουν την ρήτρα διαφύλαξη που θα ισχύει, που έχουν σήμερα και μπορούν να ακολουθήσουν την ρήτρα. Αλλά η διαδικασία αυτή περιέγραψε ο Πίτερ Λίζε. Εξετάζουμε τη ρήτρα διαφύλαξη, πάμε στην ΕΦΣΑ για να υπάρξει αξιολόγηση ότι υπάρχει πράγματι λόγος για προστασία της υγείας ή του περιβάλλοντος να γίνει χρήση της ρήτρας διαφύλαξης και αν ξανά πει ουχή η ΕΦΣΑ δεν υπάρχει ουδής κίνδυνος για το περιβάλλον για την υγεία και λόγος να χρησιμοποιηθεί ρήτρα διαφύλαξης θα πρέπει να αποσύρει αυτή τη ρήτρα το κάτω μέλος ή αλλιώς το πάμε το κράτος μέλος στο δικαστήριο. Αυτή η αλλιως το παμε το κατω μελος προβλέπεται. Δεν αφαιρούμε δικαίωμα κράτους μέλους να αμφισβητήσει και να στραφεί, να φεσιβάλει μια απόφαση για λόγους περιβαλλοντικούς ή λόγους υγείας. Προσθέτουμε στα δικαιώματά τους μια πολύ απλούστερη διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν να πούν όχι. Αυτό κάνουμε. Βεβαίως δεν εγκρίνω το να μαθαίνει κανείς από τις εφημερίδες πράγματα τα οποία θα συμφωνηθούν αύριο. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ όταν συναντιόμαι, συναντιέμαι μετά από δύο μέρες μάλλον άλλον επίτροπο. Αυτά είναι πράγματα που δεν εγκρίνουμε αυτή η διαρροή ειδήσεων στις εφημερίδες. Ο ε, κύριος Σόμες αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό θέμα που θα ήθελα να θίξω. Να μην ενημερώνονται οι καταναλωτές για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς και την καινοτομία θα έλεγα εν γέννη. Διότι διατρέχουμε τους ίδιους κινδύνους σε διάφορα μέτωπα όσον αφορά την καινοτομία στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, αλλά η διαδικασία καινοτομία. Και πραγματικά πιστεύω ότι πολλοί φορείς απουσίαζαν από τον διαφωτισμό αυτό, από την ενημέρωση ε, των καταναλωτών. Ε, όλοι φταίνε. Και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κοινοβούλιο και η ίδια βιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης, οι πάντες θα Όλοι έμειναν πίσω. Εξού και το κενό που καλύφθηκε από τις φήμες που δημιουργούσαν τρόμο. Διότι αυτή η φωνή μόνο ακουγόταν. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Μέσω στοιχείων και όχι μέσω προπαγάνδα υπέρ των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αυτό με ενδιαφέρει καθόλου, μα καθόλου. Αλλά πρέπει να δοθούν τα στοιχεία, να μιλήσουν οι επιστήμονε, να πούν ποια είναι τα στοιχεία και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει αναφερθούν στου κινδύνου. Και θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία στο τραπέζι μπροστά μα, ούτω ώστε σαν έξυπνα ανθρώπινα όντα να πάρουμε έξυπνε αποφάσει. Περί αυτού πρόκειται, λογική συζήτηση που ήδη ζητήθηκε επίσης από την κυρία Και συμφωνώ με την κυρία Συμφωνώ, την υποστηρίξω και όντως θα πρέπει να έχουμε πιο ανοιχτόμυαλες απόψεις για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα να μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας και την απόφαση της Επιτροπής. Το τα βλέπουμε πρώτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η μοίρα μας και η μοίρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα σας ξαναδούμε φυσικά αργότερα με τις επαληθεύσεις και τις νέες διαδικασίες που προτείνετε. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν με τις νέες εμπειρίες. Ευχαριστώ. Αύριο το πρωί έχουμε ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι, να είσαστε στην ώρα σας και προς το παρόν πέρασε συνεδρία σας. Χαίρετε.